Buenos días. Good morning, sirs and madams. Renaudamos, renaudamos la sesión. Συνεχίζουμε την χθεσινή συνεδρίαση και θα μας απασχολεί το σημείο 9 και 10 της μεσαίας διατάξεως, τα οποία θα εξετάσουμε ομού. Το σημείο 9 αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού 1060-2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοποιητικής ικανότητας και το σημείο 10 συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένου οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις οδηγιες 2011 2011-61 σχετικά με του διαχειριστέ οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Θα δώσω το λόγο δίχως καθυστέρηση στον εισηγητή κύριο Λεωνάρντο Ντομένιτσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω για την οργάνωση των εργασιών μας, ε, να γνωρίζουμε τους χρόνους ε, ομιλίας. Εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ σύντομο στην ε, παρουσίαση την αρχική για να αφήσω λόγο στους συναδέλφους και να ακούσω τις απόψεις τους εκ τούτου και έπειτα να κρατήσω λίγο χρόνο για μένα προκειμένου να απαντήσω στο τέλος. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι χρόνο έχουμε και έχω στη διάθεσή μου και για τις δύο εκθέσεις έχουμε μέχρι τις 10 και 30. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 10 και 30 διότι όπως γνωρίζετε θα φτάσει ανάμεσά μας ο Ούγγρος οικονομικό, ε, ε, Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, πόσο χρόνο χρειάζεστε στο τέλος προκειμένου να απαντήσετε στις παρατηρήσεις στα σχόλια. 5-6 λεπτά. Μεταξύ 5 και 7. Δεν ακούτε την διερμηνία. Ναι, ναι, όχι, τα λειτουργεί πρώτα, λειτουργεί. Παρατήρησε εκτός μικροφώνου. Έχουμε δύο θέματα που θα μας υποσχολήσουν πριν από 10 και Πρόεδρος. Θα ε, εξετάσουμε από κοινού και τα δύο αυτά ζητήματα τα 9 και τα 10 όπως είπα. Κύριε Ντομινίτσι, σας εγγυώμαι ότι 10 λεπτά πριν από το τέλος θα σας δώσω το λόγο. Θα είμαι σύντομος διότι επιθυμώ να γνωρίζω την θέση των συναδέλφων επί των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη που συνοδεύει το κείμενο. η βασική επιλογή είναι κατά πόσο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει έναν ρόλο αποκλειστικά στήριξης ή θα πρέπει να στοχεύουμε στην ενίσχυση, ενδυνάμωση κάποιων ε, σημείων που παρουσιάζονται στην έκθεση της Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο προτίθεται να κάνει νέες ε, προτάσεις, ε, νέες συστάσεις προσωπικά κρίνω πως θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δεύτερο δρόμο, δηλαδή να προσθέσουμε κάτι παραπάνω στην πρόταση της Κομισιόν. Ως εκ τούτου, καθίστε η σημερινή συνεδρίαση και όχι μόνο, θα ε, είναι, έχει μεγάλη σημασία. Ήδη έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών στο Στρασβούργο Ω εκ τούτου οι προτάσεις που κάνω ω εισηγητής είναι γνωστές και τις συνοψίζω εντάχει. Πρώτον, ένας νέος ορισμός της έννοια και της δραστηριότητας των οργανισμών αξιολόγηση. μια ε, ε, μια πρόταση σχετικά με τα δημόσιο χρέος, μια ενδυνάμωση της αρχής που περιέχεται ήδη στην πρόταση της Κομισιόν για μείωση της over-reliance, της υπέρμετρης στήριξης, του βασισμού στις, ε, στους οργανισμούς αυτούς, πλήρης ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολογήσεων σε αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων τόσο στις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των ε, οργανισμών ε, αξιολόγησης αλλά και μεταξύ αυτών και των ε, οργανισμών που που αξιολογούν Η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται στην ιδέα της ε, περιτροπής ε, που είναι κάπως περίπλοκη ε, στην εφαρμογή της, αλλά την οποία μπορώ να συμφωνήσω και προσθέτω και άλλες προτάσεις που ευνοούν το άνοιγμα της αγοράς στους αρισμούς, ουρανιούς αξιολόγησης και την πρόσβαση νέων οργανισμών, νέων οίκων μικρών στην δραστηριότητα αυτή και την ε, δυνατότητα βελτίωσης ε, των αξιολογήσεων. Επίσης ε, υπογραμμίζω το γεγονός ότι τα δημόσια χρέη, τα κρατικά χρέη, για τα κρατικά χρέη μάλλον θα πρέπει να απαγορεύεται το unsolicited, αξιολόγηση, δηλαδή αξιολόγηση που δεν έχει ζητηθεί και από πλευράς Κομισιόν ε, να συσταθεί ένας ε, ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που θα αξιολογεί τα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά κάποιες προτάσεις σχετικές με άλλες πτυχές όπως παραδείγματος χάρη το άνοιγμα της αγοράς, τη δυνατότητα πρόθεσης ε, του ε, ανταγωνισμού και το να σπάσουμε τα ολιγοπόλια, όλα αυτά περιέχουν ε, ενδείξεις και ποσοτικής φύσης, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τα ποσοστά στην αγορά, την απαγόρευση διασταυρούμενων συμμετοχών ε, όλα αυτά είναι ενδεικτικά, αλλά είναι προτάσεις που επιθυμούν να ανοίξουν τη συζήτηση και να πάνε προς την κατεύθυνση που έχει χαράξει η Κομισιόν, αλλά να προσθέσουμε νέες ιδέες και νέες προτάσεις ως Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ανταλλαγή απόψεων που μπορούμε να έχουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ ήδη από τώρα τους συναδέλφους, ειδικά τους κοιόδης ηγητάς, τον οποίων η δουλειά ήταν πολύ σημαντική και ιδιαίτερα επικοδομητική και νομίζω ότι έχουν να προσφέρουν περισσότερα. Εδώ κλείνω την σύντομη παρουσίασή μου, αφήνοντας το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Ντομενίτσι. Το λόγο τώρα έχουν οι σκιώδες ηγητές το κύριο Γκοζές από το ΕΛΚ. Παρακαλώ να βάλετε μπρος το χρονόμετρο. Θέλω να το βλέπω εκεί μπροστά μου στην οθόνη. Κάτι που μου επιτρέπει να ρυθμίσω τον ε, χρόνο μου. Πόσο χρόνο έχω, Πρόεδρε, σκιώδη ηγητές. έχετε πέντε λεπτά κύριε Γκοζές. Εντάξει, εντάξει. Σας αρκεί κύριε Γκοζές. Εγώ και με δύο λεπτά ικανοποιημένος είμαι θέλετε. Απλά θα τα πω πιο γρήγορα. Ξέρετε ότι ήμουν εισηγητής ε, τα δύο πρώτα κείμενα. Ε, κείμενα τα οποία για πρώτη φορά εισήγαγαν ε, μια ρύθμιση των λόγω οργανισμών, δημιουργώντας ένα σύστημα έγκρισης και εποπτείας ευρωπαϊκής εποπτείας. Θέλησα λοιπόν να διασφαλίσω την ε, υπηρεσία μετά την, ε, το σερβις, δηλαδή μετά την πώληση και με ιδιαίτερη λύπη είδα ότι υπήρχε αδράνεια στην εφαρμογή και οι τρεις ε, βασικοί οργανισμοί τους οποίους ακούμε καθημερινά ενεκρίθησαν το 30 Οκτωβρίου 2001 και έχουν καταθέσει τους φακέλους το Σεπτέμβριο 2010. Εξάλλου, τα κείμενα που βρίσκονται σε ισχύ τώρα δεν εφαρμόστηκαν ουσιαστικά και η εποπτεία η προγραμματισμένη δεν υλοποιήθηκε διότι φυσικά η έγκριση ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου, άρα χρειαζόταν και κάποιο χρόνο για να επαληθεύσουν κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί πληρούσαν τις προϋποθέσεις ε, τις οποίες οι ίδιες είχαν αναγγείλει. Ε, λοιπόν, ενώπιον αυτής της καταστάσεως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί και σήμερα να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν, ε, ε, έναν, έναν, ε, έναν κανονισμό πολύ λεπτομερή, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να εφαρμόσετε. Υπάρχει λοιπόν δράνει όλων των εμπλεκομένων, των ίδιων των οίκων, των επενδυτών, όσων χρησιμοποιούν αυτές, αυτές τις αξιολογήσεις, αλλά θα πρέπει να, νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση ώστε τα πράγματα να μην προχωρήσουν καθόλου. Λοιπόν, το μόνο ζήτημα για τις οίκους είναι η υπερβολική εξάρτηση από τις αξιολογήσεις των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Όπως, και αν, όπως προτείνει ο Επίτροπος, κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στα κείμενα και σταματήσουμε να προσθέτουμε νέα κείμενα, διότι το παράδοξο είναι εδώ. Θα πρέπει να υπάρξει να αποτοξίνωση από τις, από ε, τους οίκους αυτούς, γι' αυτό είμαι και υπέρ, και στα νέα κείμενα μιλάμε για τις ε, οίκους αυτούς. Λοιπόν, θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε και να ενεργούμε σχιζοφρενικά. όταν θα έχουμε ρυθμίσει λοιπόν ε, αυτή την υπερβολική ε, ε, ε, αξία αυτών των αξιολογήσεων, λοιπόν άκουσα ότι οι μη ζητηθήσει αξιολογήσει θα πρέπει να απαγορευτούν. Θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό διότι αξιολογήσει έχουμε παντού και πάντα. Όταν εγώ μιλάω, με αξιολογούν, με σημειώνουν. Και όταν δεν μιλάω πάλι και αν δεν υπάρχει μια επίσημη δημόσια αξιολόγηση, εν θα υπάρξουν ε, κάποιες ε, αξιολογήσεις ε, υπόγειες που θα... επίσης η ευθύνη των οίκων από τη στιγμή που αφαιρούμε από την οίκους αυτό είναι τον σοβαρό χαρακτήρα, πούμε, και αυτό είναι τον ιερό χαρακτήρα, θα που του έχουμε δώσει, θα μπορούσαμε λοιπόν να αποδεχτούμε από αυτέ. Τώρα, ο ρόλο ε, τη ΕΣΠΑ υπάρχει κίνδυνο ε, ότι δηλαδή θα αποδυναμωθεί η ΕΣΠΑ. Ε, κάτι αυτό δεν, αυτή η σύσταση, η ίδρυση μάλλον δεν αξιολογήθηκε από κανένα ούτε από τα κρατημέλη ούτε από τις ίδιε ε, από τους οίκους. Αυτό είναι να δημιουργείο το κοινοβουλίο και θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε από να αποδυναμώσουμε την ΕΣΜΑ και να την καταστήσουμε έναν οργανισμό δίχως ε, ευθύνες, ανεύθυνο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι φορά. Μετά ε, έχουμε να μιλήσουμε για τις συγκεντρώσει, ε, για τις αγορές κλπ. Αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η αξιολόγηση να είναι ένα στοιχείο ενημέρωσης και τίποτα παραπάνω για τους επενδυτές και για όλους όσοι συμμετέχουν στην οικονομική ζωή. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση τώρα για τα δημόσιο χρέος. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε τακτά διαστήματα και εκτός από αυτών των ημερομιών των συγκεκριμένων και σαφών δεν μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η αξιολόγηση. Ναι, εντάξει, μπορεί να προκύψει κάποιο γεγονός, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι ένα φοβερά σημαντικό γεγονό. Δεν μπορούμε καθημερινά, κάθε ώρα και στιγμή οι οίκοι να τροποποιούν τις ε, απόψεις τους ή θα πρέπει τότε να τις ε, περιφρονούμε. Τώρα, δείξαμε, όταν ε, η Γαλλία έχασε το 1α, είδαμε ότι η Γαλλία μπορούσε να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο. Άρα, μερικές φορές είναι και χρήσιμο να υποφευθούν δυο δύο-τρει φορέ τελικά δεν θα πληρώνουν καθόλου επιτόκιο. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Από την άλλη δεν υπάρχει ο σκιώδης ηγητές, ο κύριος Σμιθ, εξ ονοματός του. Πέντε λεπτά κύριε Σμιθ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά αντικαθιστώ τον κύριο Κρίντς, άρα θα πρέπει να είμαι λίγο πιο αργός. Είναι στην Ασία, κύριε Ντομίνιτζη. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας για τις ε, παρατηρήσεις σας, για τις συζητήσεις που έχουν ήδη διεξαχθεί. Αλλά ο κύριος Κλίντς θα ήθελε να ε, συνοψίσει, αν θέλετε, το συγκεκριμένες αδυναμίες ε, της, των οίκων της αξιολόγησης. Καταρχάς, η υπερβολική εξάρτηση ε, από τους ε, συμμετέχοντες της αγοράς. Ε, Ολιγοπόλια, έλεια, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, έλλειψη διαφάνειας χωρίς κοινωνική ευθύνη. Όλα αυτά αναφέρθηκαν και στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ο κύριος Κλίντς έχει και άλλες παρατηρήσεις, αλλά ξεκινάει καλωσορίζοντας τα εξή στοιχεία. Την υποστήριξη από πλευρά του εισηγητή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να περιοριστεί η υπερβολική εξάρτηση από τους παράγοντες της αγοράς. Κάποιες λεπτομέρειες ασφαλώς θα πρέπει να εξεταστούν ακόμα εισαγωγή της αρχής της ε, αναλογικότητας για τα μικρά ε, ιδρύματα πιστοληπτικής αξιολόγησης, επανεισαγωγή του MAs σε ό,τι αφορά δεκαετή περίοδο για τα μεγάλα ιδρύματα. Το θέμα είναι κατά πόσον εδώ είναι το σημείο αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων αυτών και ίσως θα έπρεπε να είναι απεριόριστο το χρονικό όριο Επίσης, αλλαγές προτείνονται στα εξή και ο κύριο Κλίντς ε, βάζει ένα ερωτηματικό εδώ. Αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα. Ο κύριος ε, Κλίντς είναι υπέρ αυτής της αρχής, όχι όμως ε, υπέρ του περιορισμού της, του μεριδίου της αγοράς. Γιατί είναι ανταπαραγωγικά αυτά που αναφέρονται για την περιορισμό του εθνικού χρέους. είναι αρχή για νέες συμβατικές εθνικές συμβάσεις δεν συνάδει με την αρχή της ε, ήπιας αξιολόγησης. Επίσης, θα ήθελε να διαγραφεί η υποχρέωση εκπεριστροφής η οποία προτείνεται. Επίσης, να διευκρινιστεί η διατύπωση σε ό,τι αφορά την έγκριση της μεθοδολογίας της ΕΣΜΑ. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν ούτε η απλοποίηση με τη βελτίωση της διαφάνειας. Και τέλος, ε, κύριε Ντομίνιτσι, ο κύριος Κλέιν σας αποστέλει εγκάρδιους χαιρετισμούς από την Ασία και προσβλέπει σε επικοδομητικές συζητήσεις τις επόμενες, τις εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί δεν εξαντλήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Κύριε Πόρτας, ε, μετά, μετά εσείς. Μετά από τους πρασίνους, ε, κύριε Φόξ, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντομινίτση για το έργο που έχει καταβάλει εδώ η ομάδα μου υποστηρίζει τις προσπάθειές σας για την αύξηση της διαφάνειας στην αγορά και επίσης υποστηρίζουμε τις προτάσεις ε, για να περιοριστεί η υπερβολική εξάρτηση των ιδρυμάτων από την αγορά. Αλλά συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Γκόζε στο παράδοξο στο οποίο αναφέρθηκε. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την υπερβολική εξάρτηση των ιδρυμάτων αυτών, γιατί εισάγουμε τέτοια μέτρα που αυξάνουν ουσιαστικά την εξάρτησή τους, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας λένε οι κυμπιστροπτικής ικανότητες ως πηγή πληροφοριών, τίποτα παραπάνω. Αυτές οι προτάσεις όμως φαίνεται ότι τις αναγάγουν σε κάτι πολύ πιο σημαντικό, όπως και ο κ. Γκοζές λοιπόν και όπως ο κ. Σμιτ. Δεν συμφωνώ για την απαγόρευση των αξιολογήσεων σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος. Αυτό είναι κλασική περίπτωση όπου κάποιοι ας πούμε επιλέγουν να μην λάβουν υπόψη να απαγορέψουν τέτοιες πιστρεπτικές αξιολογήσεις ε, όταν δεν τους αρέσουν. Αυτό μάλλον αποσταθεροποίηση θα προκαλέσει. Ακούσατε τις ανησυχίες μου σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ε, ενός νέου ε, Ιδρύματος Ευρωπαϊκού για την επιστροφική αξιολόγηση, όπως και να το ονομάσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχει όφελος στην δημιουργία μια νέα υπηρεσία, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους. Αν η, η δημιουργία ενός ε, τέτοιου Ιδρύματος θα οδηγήσει στον κόσμο να εξαρτάται από αυτό, απλά και μόνο επειδή ε, χρησιμοποιεί δημόσιου πόρου. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να μειώσει την υπερβολική εξάρτηση ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλει να βελτιώσει τον ανταγωνισμό. Ότι θέλει να μπουν νέοι φορεί ε, και νέοι παίκτε στην αγορά. Πώ θα το πετύχουν αυτό το σκοπό που είναι αξιόλογο. Χρησιμοποιώντα, δημιουργώντα ένα δημόσιο σώμα το οποίο θα είναι κατά των στόχων αυτό. Ούτε για το καθεστώ τη αστική ευθύνη μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αν ε, τεθεί, αν εφαρμοστεί η αστική ευθύνη, προφανώ οι επενδυτέ θα εξαρτούνται πιο πολύ από τι ε, αξιολογήσει των επιστρεπτικών ιδρυμάτων και θα αυξαθεί θα μειωθεί το κόστος εισαγωγής στην αγορά, θα αυξηθεί το κόστος ε, εισαγωγής στην αγορά και είμαι βέβαιος ότι τα μεγάλα επιστρεπτικά εντρήματα θα έχουν πιο πολλούς πόρους για την ε, υποχρεωτική, την εκπεριστροφή υποχρέωση. Έχω σοβαρές αμφιβολίες. Ε, τα μικρά ιδρύματα πιστροπτικής αξιολόγησης Πού πιστεύετε, που, που δρούν σε περιορισμένες ε, αγορές, πού θεωρείτε ότι θα στραφούν. Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει μια περιστροφή μεταξύ των μεγάλων παικτών για την αύξηση του ανταγωνισμού. Ευγενής στόχος της πρότασης αυτής, θεωρώ. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά πώς θα το πετύχουμε αυτό. Δεν μου αρέσει αυτή η υποχρέωση εκπεριτροπής. Αλλά θεωρώ ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε και κύριε Ντομινίτσι αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσατε να εξετάσετε κάποια άλλη μορφή αύξησης του ανταγωνισμού. Ίσως όταν μία τράπεζα ή κάποιος που εκδίδει ένα ομόλογο ή ένα οποιαδήποτε άλλο μέσο θα πρέπει να έχει παραπάνω από μία έκθεση αξιολόγησης. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μία αυτή μία από αυτές τις εκθέσεις να προέρχεται από ένα μικρό ίδρυμα πιστοληπτικής ικανότητας. Δηλαδή, να είναι ένα άλλο ίδρυμα. Όχι το Standard όχι το Moods, όχι το Finchie. Αυτή η διάταξη θα πρέπει να εξεταστεί εντελεχώς. Εγώ θα προτιμούσα να ρωτήσουμε τους μεγάλους οίκους αξιολοπτικής ικανότητας πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Μπορεί να μην θέλουν βέβαια να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αλλά αν δεν καταθέσουν κάποια αξιόλογη πρόταση θα καταλήξουμε σε αυτή την υποχρέωση εκπεριτροπής. Άρα θα τους ρωτήσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ε, σύστημα που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα τώρα σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις τριτών χωρών. Κάποιες χώρες περνούν αλλαγές στο καθεστώ του για να συνάδουν με το CRA 1. Και άλλες αλλαγές στα πλαίσια του CRA3 θεωρώ ότι θα καθυστερήσουν και μόνο αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει στο Κοινοβούλιο να βάλουμε μία τελεία, να σταματήσουμε αυτή την υπερβολική ρύθμιση, γιατί όταν τίθεται σε εφαρμογή μία νομοθεσία, αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά να επεξεργάζεται μία άλλη νομοθεσία καινούργια. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. κύριο, στον κύριο Σμίθ οφείλεται τον επιπλέον χρόνο που μιλήσατε. Ο κύριος Καφέ, ξενομέρος των Πρασίνων. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να επανέλθω στην αρχή της παρέμβασης του Ζων Πολγκοζές, ο οποίος είπε ότι πριν δεν πρέπει να έχουμε κανένα, μια ρύθμιση πολύ λεπτομεριακή. Δεν πρόκειται για κανονισμό. Τότε δεν θα πρέπει να κάνουμε ούτε για τα δημόσια ελλείμματα, ούτε για τα κράτη-μέλη, ούτε για τα διορθωτικά ελλείμματα κλπ. Συμφωνούμε, τα διαγράφουμε όλα αυτά και τώρα θα μπορούσαμε να βρούμε ένα συμβασμό, διότι δεν υπάρχει λόγος να συμπεριλάβουμε τα κράτη-μέλη σε μια εθνική πολύ λεπτομερή και αν πούμε ότι για τις οργανισμούς αξιολόγησης δεν θα πρέπει να είμαστε λεπτομεριακοί, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Δεν ε, τώρα για τους οίκους αξιολόγησης Όλοι συμφωνούμε πως ε, το πρώτο διακύβευμα είναι να περιορίσουμε την εξάρτηση των αγορών. Και αυτό, ε, αντίθετα από τον Πόρτο Γκοζέ. με το πρώτο μέρος της ομιλίας του Γκοζέ είμαι σύμφωνος. να δηλαδή, αυτή είναι προτεραιότητα υπερθυμών ένα. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσουμε τροπολογίες ώστε να συμπεριλάβουμε στο EFM και στο SITS το γεγονός ότι τα ε, οίκοι που τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις ε, δεν θα πρέπει να ε, τηρούν μια ρήτρα αυτόματη και να είναι υποχρεωμένα τα κράτη ή οι οργανισμοί να απολύσουν αν υπάρχει υποβάθμιση κλπ. Ε, θα πρέπει να έχουμε αυτή την ε, συζήτηση. Εγώ δεν είμαι διαπραγματευτής, του ΣΕΑΡΔΕ, αλλά πρέπει να έχουμε μια, συζήτηση, κύριος Γκοζές ε, δεν χρειάζεται να αυξηθεί περαιτέρω η σημασία των οίκων αξιολόγηση. Σχετικά με την εξάρτηση, προσπάθησε να περιορίσει τις ε, περιπτώσεις όπου τα κρατημένη μπορούν, τα αξιολόγηση μπορούν να μειώσουν την αξιολόγηση και την διαβάθμιση των κονδύλων. Άρα πρέπει να έχουμε κάποιε ημερομηνίε συγκεκριμένε ε, για να εκδίδουν ε, νέες αξιολογήσει εκτός από έκτακτες περιπτώσεις. Ε, τώρα, σχετικά με τη μείωση τη εξάρτηση των αξιολογήσεων, αυτό περνάει μέσα από τη μείωση των τον συμβολισμό των λέξεων. Μιλάμε για υποβάθμιση, μιλάμε για υποβάθμιση ενό ενός Εάν περνάμε από την υποβάθμιση σε ενδεχόμενα μιας ε, αδυναμίας ε, πληρωμής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αυτή η αδυναμία πληρωμής, ε, η αφαιρεγιότητα. Εάν λοιπόν οι αξιολογήσεις μας έδιναν αυτή τη διαβάθμιση, τότε δεν θα βρισκόμαστε πλέον σε μια συμβολική λογική της αξιολόγησης της κρίσης, αν θέλετε, από πλευράς ε, οίκων αξιολόγησης επί κρατών. Θα μιλάμε για αξιολόγηση σχετικά αντικειμενική μιας ε, δυνατότητας ε, αδυναμίας πληρωμών που θα γνωστοποιείται στους επενδυτές. Αυτό θα επιτρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε την εργασία των οίκων, διατηρώντας όμως τις απαραίτητες προφορίες για τους επενδυτές φυσικά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θεωρεί σημαντικό για να μειώσουμε την βαρύτητα των οίκων είναι οι προγνώσεις. Οι οίκοι χρησιμοποιούν λοιπόν δείκτες κάνουν ε, διαγνώσεις αλλά κάνουν και προβλέψεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι. όταν μιλάμε για την κεντρική τράπεζα, μιλάνε για την κεντρική τράπεζα, λέω ότι έχουν δίκιο. Όταν επικρίνουν τις πολιτικές λιτότητες λέω ότι έχουν δίκιο. Όταν θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασία, δεν συμφωνώ μαζί τους, αλλά δεν έχει σημασία αν εγώ συμφωνώ ή όχι. Το ζήτημα είναι αν αυτό είναι ο ρόλος των οίκων να κάνουν προβλέψεις για τις δημόσιες πολιτικές ο ρόλος τους είναι να δείξουν, κάνουν μια αξιολόγηση σχετικά με την φεραγιότητα ή την αφαιρεγιότητα. Εντάξει, θα πρέπει να δεσπελίσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά μόνο τη δουλειά τους και τίποτα παραπάνω. Και ε, αν έχω τα απαραίτητα δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου, να πω κάτι ακόμη, θα καλωθέσουμε τροπολογίες για να ε, συμπεριληφθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος και η μετάφρασή του για τον κίνδυνο των κρατών. Τώρα, το θέμα το πυρηνικό. Έθεσα το ερώτημα στην Moody's και το Standard Poor's και κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Είδαμε στην Ιαπωνία ότι το πυρηνικό εργοστάσιο ήταν επικίνδυνο για το δημόσιο. Άρα ο ο πολίτης πληρώνει. Λοιπόν, πώς θα λαμβάνουν υπόψη μέσω μακροπρόθεσμα αυτό το, αυτό το δηλαδή του πυρηνικού, η αξιολόγηση δεν το γνωρίζουν, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία που αξιολογούν. Εδώ δεν μιλάμε για εναρμόνιση του μοντέλου τους, αλλά θα πρέπει να τους υποχρεώσουμε να τοποθετηθούν. Και ένα τελευταίο στοιχείο Έχουμε την ε, θέση του Κοινοβουλίου στην ε, έκθεση Βόλφου Κλίντς. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά εμείς θα είμαστε υπέρ του να παραμείνουμε σε αυτήν την θέση μας ε, και να καταθέσουμε κοινέ τροπολογίες που θα μας επιτρέψουν να διευκρινίσουμε σχετικά με, το, αυτόν το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα και ποια θα είναι η μορφή του. Ευχαριστώ κύριε Καφάν. Ο κύριος Πόρτας ε, για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Γκανφάν για, τα, για τους οίκους ικανότητα, για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο πιθανότητων. Πρόκειται για θέματα και ερωτήματα τα οποία δεν προβλέπονται σε τέτοιες ε, φάσεις κρίσης. Ε, στη συζήτηση αυτή προβλήθηκαν πολλά επιχειρήματα. Αλλά το επιχείρημα του κύριου Γκόζες είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμμετέχει, αν θέλετε, στην όλη συζήτηση. Του του λεχθέντος, θεωρώ ότι μία σειρά προτάσεων του εισηγητή αποσκοπούν στην βελτίωση του συστήματος και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. σε ό,τι αφορά τα μονοπόλια, σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση της ανταγωνιστικότητας, ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του έργου των ε, οίκων πιστοληπτικής ικανότητας, ε, πιστοληπτικής αξιολόγησης. Όλες αυτές οι προτάσεις θεωρώ ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και καλό θα ήταν αν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές. Δεν ε, υποσκάπτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αυτό που κάνουν είναι να εισαγάγουν ένα πιο υγιές περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του εθνικού χρέους, προφανώς συζητούμε το θέμα αυτό εδώ σήμερα. Γιατί οι επιπτώσεις των αξιολογήσεων αυτών σε κάποια εθνικά χρέη ήταν καταστροφικές. Και γι' αυτό λοιπόν το συζητάμε αυτό σήμερα και ήταν καταστροφικές γιατί ξαφνικά αυτές οι αξιολογήσεις παρουσιάστηκαν στον τύπο με τελείως ανεξέλεγκτο τρόπο. Το ΕΛΚ και ο κύριος Γκόζες ε, προτείνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη να τίθενται υπό ε, νομική προστασία και να μην εκδίδονται τέτοιε αξιολογήσεις σε τέτοιε περιπτώσει. Αυτή η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα μεν. Αλλά μας οδηγεί σε μία επιπλέον ερώτηση, σε ένα επιπλέον ερωτηματικό. γιατί προσπαθούμε να προστατεύσουμε ένα σπίτι που έχει ήδη πιάσει φωτιά, ενώ αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μην πιάσει καν φωτιά. Και θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνέπειες της πρότασης αυτής. Θα πρέπει λοιπόν να εμπλακούμε σε πιο πρώτερη φάση, να λύσουμε το πρόβλημα πιο νωρί, όχι πιο αργά. Γι' αυτό νομίζω ότι η ερώτηση του κυρίου Καλφάν για τις πιθανότητες αποτελεί Μία καλή ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει κάτι θετικό στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία από την οποία προέρχομαι, η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι 65% και 75%. Τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει να πούμε ότι η πιθανότητα ε, χρεοκοπία στην Πορτογαλία είναι 68% και ότι η αξιολόγηση είναι β' αρνητικό. Δεν ξέρω τι πλεονέκτημα θα φέρει αυτό στο κοινό. Η, κατάσταση βρίσκεται στην... η χώρα βρίσκεται σε όποια κατάσταση βρίσκεται. Και το να πούμε ότι έχει πιθανότητες χρεοκοπίας 70% είναι θετικό. Δηλαδή, αν πουν, θα ήταν καλύτερο να λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει 98% πιθανότητες να χρεοκοπήσει. Έχω πολλές αμφιβολίες για αυτό το θέμα. Η μοναδική πραγματικά σκόπιμη λύση και λογική λύση είναι να πάυσουν οι αξιολογήσεις για τα εθνικά χρέη, γιατί εδώ εμπλέκεται ένα αντιλογικό ζήτημα, δεν πρόκειται για ένα προϊόν όπως τα υπόλοιπα. Τα ιδρύματα και οι επενδυτές το θεωρούν αυτό χρηματοοικονομικό προϊόν, αλλά σε ό,τι αφορά τους φορολογούμενους, αυτό δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύσει και άρα να μην εκδίδονται τέτοιες ε, αξιολογήσεις. Ε, αυτό ε, θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Μπορεί κανείς να έχει τη δική του προσωπική εκτίμηση, αλλά όχι επίσημη αξιολόγηση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτή είναι η μοναχική λογική απάντηση για την κρίση αυτή. Και τώρα να πω το εξή, ότι άμα να αλλάξουμε την κατάσταση θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα για το πώς θα περιοριστεί η έκδοση κάποιων ε, αξιολογήσεων. Οι περιορισμοί αυτοί θα λειτουργήσουν μόνο εφόσον υπάρχουν σαφείς νομικές κυρώσεις. Ή το σύστημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Κύριε Πόρτας, ναι, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο. Και τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τον λόγο. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφο Χουάν Τρία λεπτά. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον Λεωνάρδο για την εξαίρετη εργασία του πάνω σε αυτό το καυτό ζήτημα διότι η έκθεση αυτή εντοπίζει το σύνολο των προβλημάτων που μας απασχολούν μεταξύ αυτών είναι τα προκυκλικά φαινόμενα των αξιολογήσεων δεύτερον η, ολιγο, η δομή ολιγοπολίου που έχει δημιουργηθεί για τους αξιολόγησης και τρίτον ε, το σύγκρουση συμφερόντων. Σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα ε, η έκθεση παρέχει τις κατάλληλες και προσαρμοσμένες λύσεις. Μεταξύ αυτών των λύσεων είναι η ίδρυση ενός ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης που θα αξιολογούν πλήρη ανεξαρτησία το κρατικό χρέος ε, ο ορισμός ενός ανώτατου ποσοστού συμμετοχής στην αγορά, ενίσχυση των κανόνων που προλαμβάνουν ε, τις συγκρούσεις συμφερόντων και την απαγόρευση των ε, μη ζητησών αξιολογήσεων. Πάνω σε αυτό διεξάγεται μια ζήτηση πραγματικά σουρεαλιστική. Λοιπόν, για να ηρεμίζω κάποια πράγματα, να πω ότι υπάρχει το το ποδόσφαιρο το οποίο θα δούμε στην τηλεόραση απόψε, αλλά ό,τι και αν πιστεύουν οι οπαδοί ενώπιον της οθόνης είναι ο διαιτητής ο οποίος ε, σημειώνει και αξιολογεί. Και εδώ αυτό έχει σημασία, δηλαδή η αξιολόγηση των οίκων. Διότι η πρόταση αυτή νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη και κατάλληλη Τώρα, αν έχουμε ένα μοντέλο το οποίο ο εκδότης πληρώνει, είναι μοναδική λύση που μπορεί να είναι πιστική. Ορισμένοι εφαρμόζουν τον, ε, την αρχή επενδυτής, ε, εκδότης επενδυτής, ε, τότε η πρόταση του Ντομινίτσι είναι η μόνη δυνατή. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτές οι προτάσεις είναι αξιόπιστες και ελπίζω οι βουλευτές ε, της ε, Επιτροπής μας και οι βουλευτές του Σώματος γενικότερα θα έχουν το θάρρος να τη στηρίξουν. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά, η κυρία Βουικστρόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Εδώ στην Επιτροπή βρίσκομαι για πρώτη φορά σήμερα και γιατί, γιατί είμαι μάλιστα η συγκήτρια της ε, γνωμοδότησης ε, της σχετικής με τη σχετική έκθεση από την Επιτροπή Γιούρι. Χαίρομαι που μου δώσατε το λόγο. Αναφέρατε κάποιες από τις σκέψεις μου. Σκοπός μου είναι να σας ε, δώσω μία γνωμοδότηση που θα εστιαστεί στις βασικές αρμόδιοτητες της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά το αστικό και το εταιρικό δίκαιο και ασφαλώς το πιο σημαντικό στοιχείο θα είναι η αστική ευθύνη, η σχετική πρόταση που έλπιζα να συζητήσω εδώ σήμερα. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, όπως και εσείς εδώ στην Επιτροπή σας, έχει ζητήσει να υπάρχει ένας κανονισμός ε, κοινό για την αστική ευθύνη για του ε, οίκου πιστοληπτική αξιολόγηση. Χαίρομαι που το συζητάμε λοιπόν αυτό σήμερα, αλλά θεωρώ ότι χρήζει βελτίωση η πρόταση, η πρόταση για την αστική ευθύνη τη Επιτροπή εισάγει ένα σύστημα όπου τα μέρη θα πρέπει να διευκρινίσουν πολλά ζητήματα. Καταρχάς θα πρέπει να συζητήσουν κατά πόσον ε, υπήρξε παραβίαση του κανονισμού και κατά δεύτερον κατά πόσον η παραβίαση αυτή επηρέασε την αξιολόγηση. Για τα δύο αυτά θέματα το βάρος αυτής ευθύνης αν θέλετε το έχει ο οργανισμός πιστοληπτικής ικανότητας αξιολόγησης. Άρα ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να ε, αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του κανονισμού και ότι η ενδυνάμει παραβίαση δεν επηρέασε την αξιολόγηση. Με άλλα λόγια, ο επενδυτής και πάλι θα πρέπει να αποδείξει ότι ένας οργανισμός έλαβε μία απόφαση η οποία όμως χρήσεται ευκρίνηση τώρα για να καθοριστεί αν υπήρξε παραβίαση των κανόνων προτείνω να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη διαδικασία στα πλαίσια της ΕΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 23, πέμπτη παράγραφος του κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΜΑ διαθέτει ήδη μια διαδικασία βάσει της οποίας αποφασίσει κατά πόσον υπήρξε παραβίαση του κανονισμού ή όχι. Και η διαδικασία αυτή δύναται να καταλήξει σε πρόστιμο προς τον Οργανισμό Επιστολεπτικής Αξιολόγησης. Αυτό δεν, δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει ε, τα μέρη να αποφασίσουν κατά πόσον υπήρξε παραβίαση ή όχι. Κατά δεύτερον, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο για έναν επενδυτή να συλλέξει αποδεκτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά ε, ενδυνάμει παραβίαση η οποία οδήγησε σε λανθασμένη αξιολόγηση. Το κριτήριο και το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί ε, ένα από τα βασικά στοιχεία, μία από τις βασικές αρχές της αρχής μας και θα πρέπει και εδώ να ισχύσει. Δεν θεωρώ ότι είναι αναλογικό και σωστό να εγκαταλείψουμε την αρχή αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση και γι' αυτό λοιπόν θα προτείνω στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων το βάρος της απόδειξης να τοποθετηθεί, αν θέλετε να το φέρει ε, το μέρος που ισχυρίζεται ότι υπήρξε παραβίαση. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικές αρχές, ξέρετε, και πρόκειται για ένα σημαντικό κανονισμό. Το γεγονός ότι ήδη έχει αναθεωρηθεί τρεις φορές το αποδεικνύει αυτό. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να προασπιστώ μία λογική, αναλογική προσέγγιση με κάποια προσοχή προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καθεστώς κανονικό σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη και να αξιολογηθεί και ε, ο αντίκτυπος του μετά από κάποια χρόνια για να δούμε κατά πόσο πετύχαμε τους στόχους μας και να κλείσω λέγοντας το εξής. Κύριε Ντομίνιτσι, εισάγατε μια τροπολογία για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ό,τι αφορά το αστικό δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχω καταθέσει εγώ σχετικές τροπολογίες ακόμη, Είμαι βέβαιη ότι η Επιτροπή μας θα το συζητήσει το θέμα αυτό. Δεν είμαι πεπισμένη ότι είναι σωστό να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε κάθε νομοθέτημα όταν, πρόκειται, όταν έχουμε ε, οριζόντια εργαλεία προς αυτό το σκοπό, τα οποία λειτουργούν μια χαρά. Άρα θα σας ξαναπαρουσιάσω στην Επιτροπή σας ποιες είναι οι σκέψεις μας στα πλαίσια της δικής σας Επιτροπής και κατευθείαν Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις προσπάθειές σας και καλή τύχη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βίξον. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαν για τρία λεπτά. <clears throat> ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Συμμετείχα το Γενάρη στην ακρόαση για το θέμα των οργανισμών ε, αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα και είχαμε κάποιου πολύ συμπαθεί. Ε, ανθρώπους εδώ, αλλά το θέμα που τίθεται είναι τι μπορούν να κάνουν ο Ιάπωνας εκπρόσωπος ήταν ο μεγαλύτερο. Είπε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη. Θέλουμε να έχουμε την ευθύνη για τα στοιχεία που δίνουμε. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ε, είναι κάτι που ε, ε, δέχτηκαν όλοι. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός όχι να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε στου τρει μεγάλους όπως είπε κάποιος, αυτό ήταν κάτι που παρεμποδίστηκε μέχρι στιγμής, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή να υπάρχει ένα πεδίο νέων οργανισμών αξιολόγηση. Ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές ναι, το ακούσαμε στην ακρόαση αυτή και είπαν ότι θέλουμε να είμαστε πιο διαφανεί. θέλουμε οι μελέτε που γίνονται να περνάνε στο διαδίκτυο, να ξέρουμε ποιε ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και ποια τα αποτελέσματα στο οποίο καταλήξαμε. Μια διαφορετική ποιότητα. Ε, τώρα, πώ μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι, αυτοί οι οργανισμοί. Η μία δυνατότητα θα είναι να δώσουμε στα Ιδρύματα τη δυνατότητα εξασφάλισης της ανεξαρτησίας αυτών των οργανισμών αξιολόγησης και να, ε, ε, μπορούμε για να υπάρξει ένα οργανισμό αν κάποιο πει ότι εντάξει ιδρύω εγώ ένα τέτοιο οργανισμό, σας λέω ποιος ε, καλύπτεται κάτω από αυτό και έχω το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμή δεν γινόταν κάτι τέτοιο. Πολλοί από του συμμετέχοντε στις, οργανισμού οργανισμούς ανακαλύψαμε ποιοι είναι μονάχα όταν επέμεινε κανένας να πάρει το στοιχείο αυτό. Δεν μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μου φαίνεται κύριε Σιγητά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανένας ευθύνη για τα αποτελέσματα. Όταν λέω κάτι θα πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για αυτά που λέω. Η ε, ανεξαρτησία ή μη των ε, οργανισμών αξιολόγησης ε, θέλουμε να υπάρχει επίσης μικρότερη δυνατότητα επίδρασης ε, των οργανισμών αυτών. Εγώ ρώτησα ε, γιατί εξαρτώσαστε τόσο πολύ από τα αποτελέσματα των οργανισμών αξιολόγησης. Ε, και η απάντηση ήταν ναι, σε όλους τους τομείς υπάρχουν αυτού του τύπου οι οργανισμοί. Δεν είναι ένας παράγοντας τοσο πολλούς όπως συσχετίζονται, και γι' αυτό στο σημείο 8 λέει ότι εάν υπάρχει μείωση του, του βαθμού δεν πρέπει να οδηγήσει αυτό αυτόματα σε, ε, σε πώληση των ε, μετοχών αλλά θα πρέπει οι ε, εκδίδοντες τις μετοχές αυτές να αξιολογήσουν μόνοι τους τις, ε, ε τις ε, μετοχές αυτές. Τώρα για το, τη διατησία έχουμε το ε, ποδόσφαιρο ε, Γαλλία Γερμανία σήμερα, έχουμε το κόσμο, έχουμε το Ρίχτερ. Καμιά φορά οι διαιτητές μπορούν να κτηρούν τους, αγώνες, τους κανόνες. Αλλά θα πρέπει βέβαια να έχουν τους κανόνες στα χέρια τους για να μπορούσουμε μετά να αξιολογήσουμε. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό διατητή. Ελπίζω και οι δύο ομάδες να έχουν πολλή επιτυχία. Δεν σας πω ποια από τις δύο ομάδες προτιμώ. Ωραία, α έχουν και οι δύο ομάδες τύχη και βλέπουμε. Η κυρία Πε... τρία λεπτά παρακαλώ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Διαιτητά. Θα θυμάται ο Πολ Κοντζές ε, το 2008 όταν ήταν εισηγητής για τους οργανισμού αυτούς αξιολόγηση. Ε, είχα θέσει το, μια τροπολογία για την, μια δημόσια υπηρεσία της αξιολόγησης και είχα θέσει το θέμα του κρατικού χρέους. Εν τω μεταξύ βέβαια αυτό ο φάκελος δεν προχώρησε όσο πλευρά θέλαμε. Και λέχθη ότι δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά όχι επειδή δεν καταφέραμε να περάσει ο φόρος των χρηματοπιστικών συναλλαγών ε, έχουμε εγκαταλείψει κάθε ιδέα όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ο τέος επίτροπος Τσάνι Μακρύβη είχε πει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε οργανισμούς αξιολόγησης ε, και να το θεωρούμε ότι είναι η πηγή όποιου κακού υπάρχει στις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Ε, εντάξει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα άσχημα της ε, κρίσης, όλα τα, τα προβλήματα της κρίσης και δεν πρέπει να παραβλέψουμε λοιπόν τους οργανισμούς αυτούς. Όχι επειδή τα πράγματα δεν προχωράνε όσο γλίγορα θα θέλαμε, δεν πρέπει να δρανίσουμε, σίγουρα όχι. Δεν είναι αυτό προς τιμή του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποβάλουμε θετικές προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε την αδράνεια που φαίνεται ότι καμιά φορά διέπει την Κομισιόν. Θεωρώ ότι υπάρχουν στην έκθεση πολλά στοιχεία του Λονάδο Μινίτσι που πάνε προ την καλή κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη τροπολογία 27 στον αφορά τον τρόπο αμοιβή των ε, υπηρεσιών ή η τροπολογία 38 στον αφορά το δημόσιο χρέο. Θα ήθελα να επανέλθω στην ιδέα αυτή του ιδρύματο που συζητήσαμε στα πλαίσια της έξι πρωτοβουλίας του Βολφ Klintz. Πολλές από τις πτυχές της συζήτησης για τους οργανισμούς αξιολογήση. Ε, ξαναεπανέρχονται όταν εξετάμε τα κανόνες λογιστικής. Και μέσα στον τομέα αυτό, που είναι ο πρώτος ε, τομέας που από τη δεκαετία του γνώρισε πραγματική παγκοσμιοποίηση, εξετάστηκε η λύση του Ιδρύματος μετά από αποτελέσματα που είναι γνωστά. Δηλαδή, αυτοδιακανονισμός και ιδιωτικοποίηση ενός θέματος που είναι κατά βάση ένα κοινό αγαθό της οικονομίας να μην κάνουμε το ίδιο σφάλμα. Ε, ξέρω απόλυτα την συζήτηση που υπάρχει στη Γερμανία για μη ένα ιδιωτικό ίδρυμα. Είμαι ρα... δι... Ε, ριζικά αντίθετη γιατί θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε με τους λογιστικούς κανόνες. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σφάλμα να μην ξεχνάμε τι έγινε τότε με την ΕΣΠΕ. E τι τις κατηγορούμε ότι περνάει μόνο με την, ε, το σκεπτικό των ε, λογιστικών εταιριών των μεγάλων τεσσάρων χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλους τους άλλους. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ μιας δημόσιας ε, ε, υπηρεσίας ε, αξιολόγησης, αλλά είμαι αντίθετη κατά μιας ε, ιδιωτικής Και θα το ίδιο με εκείνο που κάναμε με την Εδώ τελειώνει κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που με επιτρέψατε να ξεπεράσω λίγο το χρόνο μου. Όχι, μην μη στεναχωριέστε κύριε Βερές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Γκυγιόλ έχει το λόγο. Ορισμένα λίγο σημεία. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Λεωνάρδο για την έκθεσή του. Έχω κάποια σύντομα σχόλια όσον αφορά το θέμα για το οποίο θα είμαι συγητής για την επόμενη αναθεώρηση. Δεν καταλαβαίνω πλήρως ίσως τις, ε, κάποιες από τις τροπολογίες σας. Γιατί προτείνετε να διαγραφεί η αυτόματη χρήση των ε, οργανισμών αξιολόγησης. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι έχετε κατά νου για τη συζήτηση για του οργανισμού αξιολόγηση, ένα από τα κύρια θέματα για μένα είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών ε, παραγόντων. Για τους μεγάλους δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα να αξιολογούνται τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στα οποία ήδη επενδύουν. Και εκεί θα έλεγα δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει μια αναφορά και μάλιστα μια αυτόματη αναφορά στις υπηρεσίες ε, αξιολόγησης χρηματοληπτικής ικανότητας άμα δίνουν ε, δηλαδή χρήματα σε μικρές εταιρείες ε, τις αξιολογούν εκείνοι αν δίνουν για κάποια προϊόντα θα πρέπει να αξιολογήσουν μόνοι τους πάλι θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διάκριση μεταξύ των μεγάλων και των μικρών θα είχε νόημα κάτι τέτοιο αλλά για τους μεγάλους οπωσδήποτε, δεν βλέπω γιατί στις ε, κατευθυντικές γραμμές επένδυσης για τους χρήστες, το ίδιο για τους τράπεζες κλπ, για τους μεγάλους λέω παίκτες, γιατί θα πρέπει να έχουμε αναφορά σε κάτι τέτοιο. Και παρόλο που ίσως οι μικροί παίκτες δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρως να αξιολογήσουν όλους τους παράγοντες, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε τη διάκριση μεταξύ των μεγάλων και των μικρών. Το άλλο όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγηση ε, και θέλω να σχολιάσω κάτι που είπε η Περβόν Σπυρές. Ε, υπάρχουν δύο δυνατότητες να προσφέρει κανένα ένα δημόσιο αγαθό. Μπορεί να γίνεται από το κράτος, δημόσιο δηλαδή, ή μπορεί να υπάρχει κάποιος τρίτος ε, παίκτης στον η ISP συμφωνώ ήταν ιδιωτικοποίηση του κανονισμού προς τους ίδιους τους παίκτες. Δηλαδή, οι μεγάλες τράπεζες κάνουν του δικού κανόνε, ε, τι θα πρέπει να κάνουν. Ε, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Εμεί μιλάμε εδώ για ένα ίδρυμα του οποίου ηγούνται μόνο, μόνο παίκτες απόλυτα ανεξάρτητοι από εκείνους του οποίου αξιολογούν και για τους οποίους ορίζουν τους κανόνες. Αυτό θα ήταν ίσως καλή λύση, διότι αν έχετε τα κράτη που κάνουν τους κανόνες, δημόσια δηλαδή υπηρεσία αξιολόγησης, το πρόβλημα θα είναι ότι θα υπάρχει ο κίνδυνος πολιτικής πίεσης, ούτω ώστε κάποιες υπηρεσίες, κάποιες επιχειρήσεις να είναι κάτω από πιο ευνοϊκό, ευνοϊκή αξιολόγηση. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ ενό καλά σχεδιασμένου οργανισμού, ιδρύματος μάλλον, αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκιγκούλτ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ρόχιο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα της, ε, των οργανισμών αξιολόγησης επιστολεπτικής ικανότητας, δεν θέλω να προσθέσω πολλά πάνω σε αυτά που είπε ο κ. Ντομενίτσι. Θα ήθελα καταρχήν να τον συγχαρώ για το έργο του. Ε, το πρόβλημα που έχουμε είναι η έλλειψη διαφάνειας ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά και του γεγονότος ότι επικρατούν τρεις μεγάλες ε, ε, τρεις μεγάλοι οργανισμοί σε αυτό το τομέα. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε οι οργανισμοί αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και τίποτα άλλο, να δίνουν δηλαδή ε, ε, πληροφορίες προς τους Μία ολόκληρη σειρά όρων έχουν ήδη καθοριστεί που οδήγησαν στην υπερβολική αυτή εξάρτηση, την υπερβολική εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση. Αυτό είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Έχω τέσσερις παρατηρήσεις να κάνω. Παραδείγματο χάρη το θέμα των ε, γη των ποσοστώσεων και της τη αγοράς ε, ξέρουμε ότι το γεγονός ότι κάποια επιχείρηση κινείται προς μία αλφα κατεύθυνση δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα αντίθετη με, τον κοινοτικό, με τους κοινοτικούς κανονισμούς. ξέρω ότι δεν ε, έχουμε πάντα ποσοστώσεις στην νομοθεσία μας, αλλά θα μπορούσαμε να φροντίσουμε οι μικρές ε, οι μικροί οργανισμοί αξιολόγησης να ενωθούν σε ένα δίκτυο. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο ανταγωνισμό νομίζω της αγοράς. Όσον αφορά τους μετόχους, νομίζω ότι η έκθεση πάει πιο μακριά από τη η ίδια η πρόταση της Κομισιόν. Πώς μπορούμε να συσχετίσουμε δηλαδή αυτό το θέμα με την εφαρμογή του κανονισμού που θα πρέπει να εφαρμοστεί στις, ε, ε, στους οργανισμούς αξιολόγησης σχετικά με το κρατικό χρέος. Τι γίνεται στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πελάτες των οργανισμών αξιολόγησης αν δεν έχουν δώσει την άδεια να γίνει κάτι τέτοιο και αν δεν λάβουν υπόψη το αποτέλεσμα τι θα γίνει. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας. Μετά, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης, μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε έναν οργανισμό που ίσως πέσει τελικά ε, θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Μήπως θα ήταν καλύτερη ιδέα να έχουμε έναν οργανισμό χρέους που να δίνει αντικειμενικές πληροφορίες ε, όσον αφορά το χρέος στα διάφορα κράτη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Φερέρα. για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Λεωνάρδο για την εξαιρετική του εργασία. Και θα ήθελα να τονίσω πως ε, αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Εξάλλου είναι η τρίτη προσπάθεια που κάνουμε ώστε να κατορθώσουμε να πετύχουμε κάτι και αναφίβολα θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω αυτή τη νέα πρόταση για να καταλήξουμε σε ένα σε μια απόφαση που θα είναι και υποθητή. Αναφίβολα μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση, αλλά στα βασικά στοιχεία της είναι καινοτόμος, σοβαρή και ιδιαίτερα ισορροπημένη. Υπάρχουν μερικά προβλήματα. Καταρχήν, ε, αντιμετωπίζουμε ένα ολιγοπόλιο το οποίο εγγίζει τα όρια του μονοπωλίου και το οποίο τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την ε, αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εδρυμάτων και έχει ένα πρόβλημα σημαντικό για το κρατικό χρέος, χρέος της ζώνης ευρώ. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Επί του ζητήματος ε, να πω πως το ότι ξεκινάμε από το μονοπόλιο ή λιγοπόλιο αν θέλετε που υπάρχει αποφεύγοντας ε, τις ε, διασταυρούμενες ε, συμμετοχές εδώ θα πρέπει να δούμε τις, τα ποσοστά των αγορών και όπως ακούσαμε η δεσπόζουσα θέση είναι προφανής για τους οίκους αξιολόγησης. Εδώ είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει να μελετήσουμε τις προτάσεις σχετικά με το κρατικό χρέος ε, πιο αναλυτικά. Όπως είπε ο κύριος Κοφέ, συμφωνώ με τις αναλύσεις ε, μεν, αλλά για το κρατικό χρέος ε, η δυνατότητα η πιθανότητα μάλλον αφαιρεγγιότητας ενός κράτους α, σχετίζεται με τη, από τις αξιολογήσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας φαύλος κύκλος αν θέλετε ένας παύλος κύκλος ο οποίος ε, δεν ε, ε, μας οδηγεί σε καμία λύση του προβλήματος. Γι' αυτό λοιπόν το, η ζώνη ευρώ βρέθηκε υπό την απειλή της διάλυσης. Πρέπει να δούμε το θέμα στα σοβαρά και με θάρρος. Χρειάζεται φυσικά να εξετάσουμε και τις νομικές επιπτώσεις ορισμένων προτάσεων που έχουμε εδώ. διότι δεν ε, βλέπουμε πολύ καλά πώς η λειτουργία των οίκων αξιολόγησης γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η Ευρώπη έχει ανάγκη να χαράξει το δρόμο της ε, και πρέπει να δούμε την ε, λογική αυτής της νομοθεσίας που αποφασίζουμε και τις επιπτώσεις που θα έχουν στους μικρές, στους μικρούς οίκους αξιολόγησης. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ιδέες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες η εργασία είναι εξαιρετική του συναδέλφου. Πρέπει να βελτιώσουμε τους του ε, προσανατολισμούς, αλλά το κείμενο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για σωστά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να μιλήσω και εγώ, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κάποια ομοφωνία ότι οι ίδιοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους, όπως είπε ο κύριος Γκοζές, ειδικά με το θέμα της ε, μείωσης ε, της ε, γαλλικής του γαλλικού κράτους, της αξιολόγησης του γαλλικού κράτους. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση, εξάρτησή μας από τους ε, οργανισμούς αξιολόγησης. Επίσης αναφέρουμε ότι καλό είναι να υπάρξουν νέες ε, νέοι οίκοι, αλλά αυτό εμένα μου προκαλεί κάποια σύγχυση, διότι αφενός λέμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης χάνουν αξιοπιστία και ενώ από την άλλη μεριά θέλαμε να είναι πιο ε, να δημιουργήσουμε νέους ε, οίκους, αλλά πώς ε, θα πετύχουμε αυτοί οι νέοι οίκοι αξιολόγησης θα έχουν την απαραίτητη αξιοπιστία, κάτι το οποίο χάνουν οι οίκοι αξιολόγησης που λειτουργούν τώρα. Θα δώσω το λόγο για λίγο στην Κομισιόν και μετά ο κύριος Ντομινίτση για την τελική του παρέμβαση. Ο κύριος Μάικλ Φρίντριχ ε, από την Κομισιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο Μάικλ Φρίντριχ πρόκειται να παραστεί, πάντως ε, να πω ότι εμείς εξετάσαμε την έκθεση και η θέση μας ε, βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση θεωρούμε ότι δεν είναι προς τη κατεύθυνση και εντοπίζει ο Συγητή ε, τα προβλήματα τα οποία είχαμε εντοπίσει και εμείς, θέματα εξαρτήσει ε, από του οίκου αξιολόγηση, ε, θέμα ικανότητας, αξιοπιστίας, κυρίαρχο, μάλλον συγγνώμη, κρατικό χρέος και το ζήτημα της αστικής ευθύνης. στι περισσότερε περιπτώσει ο συγητής προτείνει λύσει που πάνε μακρύτερα από τις αρχικά προτινόμενες από την Κομισιόν. Ε, το θεωρούμε θετικό αυτό. Νομίζουμε ότι η συζήτηση είναι σωστή, απαραίτητη, αν επιθυμούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Κατά τη γνώμη μας ε, υπάρχουν πτυχές που θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Το ζήτημα της εξάρτησης ε, είναι θεμελιώδες, το ζήτημα της ικανότητας είναι απαραίτητο και αυτό. Θέλουμε μια αγορά που να λειτουργεί αποτελεσματικά, θέλουμε να υπάρχουν ε, περισσότεροι οργανισμοί αξιολόγησης ε, από το ισχύον ολιγοπόλιο και ως εκ τούτου η Κομισιόν είναι της άποψης ε, πως θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο ομού με το Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Φορνιέ. Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση, αλλά με είχαν ενημερώσει ότι ο κύριος Φρίντριχ ε, θα παρίσταται από πλευρά Κομισιόν. Τέλος, ε, το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Ντομενίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους ε, για τα θετικά του σχόλια αλλά και για τις παρατηρήσεις τους. Όπως ε, είπε προλίγου η κυρία Φερέιρα, πρόκειται για ε, περίπλοκη και δύσκολη δουλειά. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε κάποιες στοιχείες. Ως εκ τούτου χρειάζεται να μπούμε στις λεπτομέρειες, ε, διότι πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο στόχος ε, επίτευξης αποτελεσμάτων μερικές φορές ε, παράγει κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα τα οποία χρειάζεται ευλόγως να ληφθούν υπόψη ε, και δεόντως, διότι με μια πρόταση προτιθέμεθα να καταλήξουμε σε κάποιο συμπεράσμα, αλλά το ζήτημα είναι τόσο περίπλοκο, ώστε μπορεί να υπάρξουν παράπλευρες επιπτώσεις επιθυμητές, μη εισελημένες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η οίκοι αξιολόγησης κάτι τέτοιο συχνά δεν το σκέφτονται και δεν το πράττουν. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν, το θέμα του κρατικού χρέους. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Θεωρώ πως σήμερα δεν θα συζητούσαμε εκ νέου για τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια το ζήτημα των οίκων αξιολόγηση εάν δεν είχε προκύψει το ζήτημα της αξιολόγησης ε, του κρατικού χρέους. Αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, αλλά είναι μια πτυχή που πρέπει να εξετάσουμε. Ως εκ τούτου χρειάζεται να βρούμε νέες απαντήσεις, νέες λύσεις διότι δεν θα έπρεπε να είναι δυνατόν για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητάει τη μη αξιολόγησή του από έναν οργανισμό αξιολόγησης. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, θέμα ευθύνης. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ε, την ιδιαιτερότητα. Συμφωνώ επ' αυτού με τον κύριο Πόρτας της αξιολόγησης ενός ε, κρατικού χρέους ε, σε σχέση με την αξιολόγηση ενός ε, ιδιώτη εκδότη ή ενός δομημένου προϊόντος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη διαφορά, διότι που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχει έναν ε, ε, αντίκτυπο και να τη κάνει αναγνώριση ε, από πλευρά νομοθεσία. Τίποτα φυσικά δεν απαγορεύει ένα κράτο να μπορεί να ζητάει να αξιολογηθεί και από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε το ζήτημα όχι μόνο από αφηρημένη σκοπιάς, αλλά και από πρακτικής σκοπιάς διότι κρίνω πως ουδής ε, κρίνει πως ε, ομολογίες που εκδίδονται από κάποια κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενέχουν κάποιους κινδύνους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Για ποιο λόγο εάν εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ε, μορφές εσωτερικής αξιολόγησης δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ενιαία οντότητα μπορεί να αποκτήσει ένα δικό της εργαλείο αξιολόγησης ε, σχετικά με την φεργιότητα του κρατικού χρέους ή όπως είπε και ο συνάδελφος η δυνατότητα εξέτασης ε, του χρέους από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής κανότητας. Θεωρώ όμως προσωπικά ότι αυτό είναι συνεπές ε, με τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Six pack, δηλαδή οικονομική διακυβέρνηση, ε, δημοσιονομικό πακέτο κλπ. Να έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του πακέτου ένα εργαλείο, να μέσο αξιολόγησης αναφορικά με την φερεγγιότητα και άρα με την κατάσταση του κρατικού χρέους των κρατών μελών εξάλλου. Έχουμε ήδη έναν οργανισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, α, θα μπορούσαμε όμως να ιδρύσουμε και μια οντότητα ex novo και να προτείνουμε διαφορετικά κριτήρια από πλευράς ε, μεθοδολογίας και αξιολόγησης όπως πρότεινε ο συνάδελφος ε, Καμπέν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα μέσο αξιολόγησης, ειδικά με την ε, πιστοληπτική ικανότητα των κρατών μελών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προσθεθεί, να συμπληρώσει τα ήδη υφιστάμενα ε, όργανα μικρών ή μεγάλων ε, οίκων αξιολόγησης. Θα ήθελα να πω επίσης πως ε, αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Γκοζές αναφορικά με την απώλεια αξιοπιστίας ε, των οίκων Αυτό είναι γεγονός, είναι αλήθεια. Αλλά το παράδοξο το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το εξής. Σε αυτή την απώλεια αξιοπιστίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται ένα αυτό με το αποτέλεσμα και μια σειρά επιπτώσεων που είναι πολύ σοβαρές από πλευράς συνολικής λειτουργίας του συστήματος. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου και ο συνάδελφος Γκίγκολντ μιλούσε για μικρές ε, οικονομικές εντότητες. Ε, λοιπόν, αν, μια, τραπεζι ένα πιστοτικό ίδρυμα ή μια οικονομική εντότητα δεν ε, έχει μια αξιολόγηση, δεν έχει αξιολογηθεί, τότε αυτόματα της ε, χορηγείται η πιο χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν ε, συμβατικές ρήτρε ε, που προβλέπουν την αυτόματη απόρριψη τίτλων σε μείωση τις πιστοληπτικές ικανότητες. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα, υπάρχει, χορηγείται τη δυνατότητα λοιπόν για την ε, εξόφληση κάποιων ε, ομολόγων σε περίπτωση που ε, η αντευτόματη ε, αυτή αποπληρωμή ε, τώρα, όπως είπε ο Γκουικλού, εγώ συμφωνώ να συμπεριλάβουμε κανόνες ε, οι οποίοι θα κάνουν διάκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων οντοτήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μετά από τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων θα ήθελα να ολοκληρώσω με δύο παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Φέγιο ότι δηλαδή χρειάζεται να συζητήσουμε σχετικά με τη σκοπιμότητα της χρησιμοποίησης του περιορισμού των ποσοστών συμμετοχής στην αγορά, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς μεταξύ μας. Ειλικρινείς όλοι συμφωνούμε με την αναγκαιότητα διεύθυνσης της αγοράς και ε, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τα μέσα για να το πετύχουμε αυτό είναι γνωστά. Είτε βρισκόμαστε στην... ακολουθούμε τη λογική μάλλον της Κομισιόν ε, αυτό, της εκπεριτροπής που μπορεί να απλουστευτεί, να τροποποιηθεί και να αλλάχθει σχετικά με την ε, περίοδο της περιτροπής κλπ. Είτε παραμένουμε στην λογική του περιορισμού των ποσοστών συμμετοχής στην αγορά ή θα εργαστούμε σε ένα εναλλακτικό πρότυπο πληρωμή ή στο συνδυασμό προτύπων, ε, μοντέλων μεταξύ του μοντέλου που βασίζεται στους εκδότες ή στο investor based model που βασίζεται στους ε, επενδυτές. Δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές. Εάν θέλουμε να ε, βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, ας βρούμε το καταλληλότερο μέσο, αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα συνδυασμό των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν υπάρχουν όμως και άλλες ιδέες, πολύ ωραία. Ευχαρίστω ε, να τις ακούσω. Αλλά χονδρικά αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Και τέλος, σε σχέση με τα όσα έλεγε ο συνάδελφος Φέγιο, ναι, είναι γεγονό ότι πρότεινα κάποιες ε, τροπολογίες ε, λίγο πιο περιοριστικού χαρακτήρα και ότι αφορά τις ε, ε συμμετοχές αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο διότι εμείς βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς και σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων αλλά πρέπει να επέμβουμε. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Καταλαβαίνω τις παρατηρήσεις που έκαναν ορισμένοι συνάδελφοι. Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων και σε ό,τι αφορά την δράση του δημόσιου τομέα πολιτικές πιέσεις και επιρροές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην, ε, κάποιες εκτιμήσεις ε, σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των κρατομελών μελών κλπ αλλά το ζήτημα είναι ότι εμεί σήμερα βρισκόμαστε σε κατάσταση σύγκρουση συμφερόνων που θα πρέπει να διευθετηθεί και σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστούμε την αρχή ότι στο σύστημα των ε, δημόσιων οργάνων και θεσμών μπορούν να υπάρχουν αυτόνομοι θεσμοί, αυτόνομοι φορεί και ανεξάρτητοι που δεν ή δεν, ε, εμπίπτουν σε, δεν υποκύπτουν σε πιέσεις ε, και άρα δεν δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων. Εγώ ε, προέρχομαι από μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών της, αλλά υπάρχουν ορισμένα θεσμικά όργανα ρυθμιστικά όπως η Τράπεζα της Ιταλίας που ευτυχώς υπάρχει και διαδραματίζει έναν αυτόνομο και ανεξάρτητο ρόλο στο πλαίσιο του θεσμικού μα συστήματος. Και αν εγώ έθετα να αμφιβάλλω αυτή την αρχή τη ανεξαρτησία και τη αυτονομία, θα αφισβητούσα συνάμα και τον ρόλο και το έργο ενός θεσμικού οργάνου που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το, οικο, το οικονομικό σύστημα της χώρας μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομινίτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατά τροπολογιών είναι 22 Μαρτίου, η συζήτηση επί των τροπολογιών στην Επιτροπή μας θα είναι 24 Απριλίου και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 21 Μαΐου. Να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική διαχείριση του χρόνου που είχαμε, διότι ακριβώς φτάσαμε στις 10.30 όπω όπως είχε προγραμματιστεί. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως.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

Okay, could, could everybody sit down, please? Παρακαλώ, καθίστε. And we, we now will proceed to the next agenda. Για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της μερικής διάταξης. So please, uh, conversations should cease. I battle with other people. Παρακαλώ, αν θέλετε να τελειώνετε τις κουβέντες σας για να συνεχίσουμε. Okay, if you could take your seats, if you're leaving, can you leave? Παρακαλώ, καθίστε ή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 Okay, Ωραία. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 11. Είναι ο οικονομικός διάλογος με την Ουγγαρία. Um, oh, <laughs> με, και ανταλλαγή απόψεων με τον ε, αρμόδιο υφυπουργό για τη στρατηγική πολιτική. Ε, ξέρω, έρχεται λίγο καθυστερημένο αυτό το θέμα, αλλά θα συζητήσουμε τη στρατηγική του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας. Ήθελα να σας θυμίσω ότι αυτός ο οικονομικός διάλογος είναι κάτι το οποίο είχαμε συμφωνήσει στο νομοθετικό πακέτο των έξι πτυχών και είχαμε έξι τομέων μάλλον, είχαμε προσκαλέσει έξι υπουργού που δεν ήταν υποχρεωτικό να έρθει, όμως αυτός ο υπουργό σήμερα δέχτηκε να έρθει και είναι ο, ο πρώτος γύρος των οικονομικών διαλόγων που θα διεξάγουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ λοιπόν ε, την ε, παρουσία. Τον ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία του. Ελπίζω να είναι μια επικοδομητική συζήτηση γιατί θα συζητήσουμε για θέματα οικονομικά. Προφανώς στην Επιτροπή που συζητάμε οικονομικά θέματα τώρα. Και θα ήθελα να του διαθέσω 10 λεπτά, έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του για να ε, μας εκφράσει τις ε, απόψεις του και εν συνεχεία θα έχουμε ένα διάστημα ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ, ε, κάντε ένα σήμα στη γραμματεία αν θέλετε να, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να συμμετάσχετε στο διάλογο με το. Και δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ να συζητήσω λεπτομερό στην οικονομική πολιτική της Ουγγαρίας. Δεδομένου ότι το προηγούμενο εξάμεινο είχαμε την Ουγγρική Προεδρία, ήταν μια Προεδρία πολύ φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι αυτό το πακέτο των έξι τομέων εισήχθη μετά την πρωτοβουλία της Ουγγαρίας και τώρα η Ουγγαρία έχει την ευκαιρία να επιδείξει την φιλική στάση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναπτύξει έναν οικονομικό διάλογο μέσα στα πλαίσια της νέας οικονομικής διακυβέρνησης. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες περνάνε πολύ δύσκολες μέρες αυτή τη στιγμή, η οικονομική πολιτική δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε μια ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά απαιτεί και μέτρα εφαρμοστικά, απαιτεί οι θεωρίες να γίνουν πράξεις και σε πολλές περιπτώσεις ε, κρατικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό στην εισήγησή μου σήμερα θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην πολιτική της Ουγγαρίας, στις πρόσφατες πολιτικές, σε συνεχεία στην εμπειρία και στα μαθήματα που πήραμε από την κρίση αυτή και, την, και τέλος θα σας παρουσιάσω την μετα, μεταρρυθμιστική μας ατζέντα. Όταν γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλωσορίσαμε τα μέτρα, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρμοστήκαμε δεδομένου ότι είχαμε ήδη μια πολύ ανοιχτή οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές. Όμως, ήμασταν και ευάλωτοι, ευάλωτοι σε εξωτερικές κρίσεις και επιρροές. Αυτή τη στιγμή το, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ουγγρικής οικονομίας είναι η αβεβαιότητα. Τίποτα δεν είναι βέβαιο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο άμεσο μέλος. Ορισμένες χώρες επισημούν μία ε, ε, ολοκλήρωση δημοσιονομική, άλλες χώρες όχι είναι σαφές ότι οι αγορές είναι ανήσυχες και ανυπόμονες με την τρέχουσα κατάσταση στις αγορές η οποία είναι αστάσμητη. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια ευρωπαϊκή κρίση, Πέρσι την Άνοιξη προσεγγίσαμε την Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή και το Δούνου του ε, για να συζητήσουμε μαζί τους ε, τα πρόσθετα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ε, το πρόβλημά μας δεν είναι η ρευστότητα, το πρόβλημά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ε, άμυνας ε, και να προβλέψουμε τους, τους ζωφερούς καιρούς και τι πρέπει να κάνουμε. όλα αυτά και να αναπτύξουμε ένα δίκτυο μέτρων για να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη της ουγγρικής οικονομίας όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να αναπτύξει ένα δίκτυο χρηματοδοτήσεων έχει καλές. Αλλά πρέπει να ε, υποστηρίξουμε και μη ευρωπαϊκές ε, χώρες και γι' αυτό η, η Ουγγαρία έχει οθετήσει ε, λίγα κατάλληλα μέτρα για να επιβιώσει. Ε, όπως ε, είχε πει παλιά ο Δαρβίνος, ε, ο, πιο ικανός θα επιβιώσει. Αλλά αυτή τη στιγμή ισχύει το ότι ο πιο δυνατός, ο πιο ισχυρός επιβιώνει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δράσουμε προληπτικά. 350 νέα νομοσχέδια έχουμε παρουσιάσει, είχαμε παρουσιάσει από το 2010 και πέρα, τα οποία καλύπτουν μια ευρία γκάμα οικονομικών στρατηγικών. Ο στόχος αυτών των νέων ε, νομοσχεδίων είναι να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ουγγαρία. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη είναι μηδενική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ουγγαρία φέτος, ε, αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα, τα προβλήματα του υπρολογισμού μας απλώς με συνεχή χρηματοδότηση. Πρέπει να αφενός να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και αφετέρου την ανάπτυξη. Γι' αυτό πέρσι η ουγγρική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,7% πολύ παραπάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο που όπως είπαμε ήταν 0, κάτι η Κριστίν Λαγκάρτ ε, του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πρέπει δημοσιονομικά, ε, δημοσιονομικές λύσεις να εφαρμόζονται με, με, λογική, με, με σύνεση και με κοινωνικό προσανατολισμό. Άρα λοιπόν είναι σωστό ότι η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς είναι ένα απαραίτητο μέτρο για την αναζωογόνηση της Ευρώπης. Το τρίτο μάθημα που λάβαμε είναι ότι πρέπει να ε, συμμεριζόμαστε και να σηκώνουμε ισομερό τα βάρη μεταξύ μας. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζονται αυτή τη στιγμή εξωτερικά και εσωτερικά με αυτές τις προκλήσεις. Ο Νίλ Φέργισον, ο ιστορικός του Χάρβαρτ, είπε ότι ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης στον ανταγωνιστικό κόσμο είναι τα διαφορετικά μοντέλα ε, που, οικονομικά και κοινωνικά. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των μοντέλων αυτών. Η, η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα συναλλαγματικά της αποθέματα, όπως το είχε επιβεβαιώσει και το περιοδικό Economist. Από την εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μία λύση η οποία να ικανοποιεί όλους. Και το δημόσιο τομέα και τις τράπεζες. Γι' αυτό ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μία συμφωνία ή μάλλον συμφωνήσουμε με τις τράπεζες μας πέρσι το Δεκέμβριο. Και είπαμε ότι στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής θα υπάρχει ισοκατανομή των βαρών θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν με τα, με μεταξύ του νομίσματός μας και των άλλων νομισμάτων και του ευρώ και ε, γι' αυτό προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε προσαρμοστικά μέτρα. Από 54 της 100 ε, το ποσοστό του κόμματός μας, ε, της, το, το ποσοστό του ελλείμματος του ΑΕΠ ήταν, ε, όταν δεν είμαστε εμείς στη κυβέρνηση, εξαιρετικά σημαντικό και η κυβέρνηση εισήγαγε ένα ειδικό μέτρο φορολόγησης των τραπεζών για να μπορέσει να εξισορροπήσει το πολύ αρνητικό ε, έλλειμμα του ισοζυγίου και να προλάβουμε περαιτέρω επιδείνωση της ύφεσης. Ε, αυτό το έλλειμμα του ΑΕΠ είχε πάει όταν εμεί δεν ήμασταν στην εξουσία από το 54% στο 80%. Ε, πρέπει τώρα το 2012 να μειώσουμε το έλλειμμα, το δημόσιο έλλειμμα από το 85% ή 82% κάτω του 80% το, το 2012. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες έντονες να μειωθεί το δημόσιο έλλειμμα και επίσης ε, το, το έλλειμμα του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Η ανάπτυξη από 6,8% που ήταν στην Ουγγαρία το 2009 ε, και μετά τη μεγάλη πτώση που σημείωσε βρίσκεται πάλι σε ανωδική πορεία. της 1η Ιανουαρίου 2013 θα εφαρμόσουμε πλέον έκτακτα μέτρα φορολόγησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο έκτακτος, η έκτακτη δηλαδή φορολογία. Τι είχαμε εφαρμόσει αυτό το φόρο για τρία χρόνια. 2009 ε, 2011 ε, και επειδή είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας και στο λόγο μας δεν θα υπάρχει άλλη τέτοια φορολόγηση. Αυτά τα προσωρινά μέτρα που είχαμε εφαρμόσει ε, χρησιμεύσαν σαν ένα, ένα τεστ δηλαδή ικανότητος για να δούμε πώς θα αναδιαρθρώσουμε, πώς θα διαμορφώσουμε τις διαθροτικές μας μεταρρυθμίσεις τώρα έχουμε υπόψη να αυξήσουμε το συνταξιοδοτικό όριο, να και να εφαρμόσουμε άλλα, μέτρα τα οποία ε, θα μας βγάλουν από την κατάσταση ενός νηπιαγωγείου που μας έχουν κατηγορήσει από γερμανικής πλευράς ε, και θα μας ενηλικιώσουν. Κατά κάποιο τρόπο σε πολλά στοιχεία η Ουγγαρία βρίσκεται στην ε, εμπροστοφυλακή άλλων χωρών ε, και προηγείται στα επιτεύγματα από ένα-δύο χρόνια. Μία, ένα από τα στοιχεία της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντα είναι να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης. Θέλουμε να, ξα, να ενσωματωθούν και πάλι στην αγορά εργασίας μακροχρόνια άνεργοι και να μην εξαρτώνται από επικρατικά επιδόματα. Έχουμε ενισχύσει τα ε, προγράμματα κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, τα προγράμματα εκπαίδευσης και η η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τομέα στην ε, ε, Ουγγαρία είναι, ε, τα συμβάλλει πολύ στην μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Και επίσης θα συνδέσουμε τις συντάξεις με τους ρυθμούς του πληθωρισμού. Άλλα μέτρα που έχουμε εφαρμόσει είναι να μειώσουμε τον εταιρικό φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 19% στο 10%, μείωση της γραφειοκρατίας η οποία ταλάνιζε τις επιχειρήσεις στην Ουγγαρία, εφαρμογή ενός φόρου κατά απόκοπήν 16% στις επιχειρήσεις Επίσης την διεύρυνση της φορολογικής βάσης ε, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν τις φορολόγησης οι μισθοί Γι' αυτό πιστεύουμε για την καταπολέμηση της διαφυγής, ότι εφαρμόζοντας έναν ενιαίο φόρο, ένα καταποκοπή φόρο θα μπορέσουμε να, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και να μην μας διαφεύγουν ε, φορολογούμενα ποσά. Ένα άλλο κεντρικό σημείο της στρατηγικής μας είναι η αναθεώρηση της, ε, της, ε, του δημοσίου, της ε, δομής του, του, των δημοσίων υπηρεσιών. Πέρσι την Άνοιξη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως σας είπα, όπου το ΑΕΠ θα βελτιωθεί κατά 2 με 3% 2012-2013 και διαθέσαμε 900 εκατομμύρια φιωρίνια ε, για την αναθεώρηση του συνταξιδοτικού τομέα. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Κόμισιον, ε, προβλέπει ότι μόνο το ίμιση των μέτρων αυτών θα εφαρμοστούν, αλλά το 2012 ήδη πάνω από το 20% των μέτρων αυτών έχουν εφαρμοστεί. Παρόλο λοιπόν που η πρόβλεψη είναι ότι μόνο τα μισά θα εφαρμοστούν λόγω εφαρμοστικών δυσκολιών, έχουμε ήδη εφαρμόσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το 2012. Και για το 2013 τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν είναι λιγότερο, που υπολείπονται από 17%. Όπως σας είπα, σε ορισμένου τομεί η Ουγγαρία προηγείται άλλων χωρών, π.χ. στην συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. την, σε πολλούς άλλους τομείς, όπως την αγορά εργασίας, η Ουγγαρία συμβαδίζει με άλλες χώρες. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος βασανίζεται με, με αυτό το πρόβλημα της απασχόλησης. Και εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στις δημόσιες μεταφορές και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως θα έλεγα ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που θα ξαναδώσουν, ε, ε, θα αναζωογονήσουν την ε, ουγγρική οικονομία. Πιστεύουμε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα αυξήσουν το ποσοστό ανάπτυξης της Ουγγαρίας και φέτος και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα κατά σειρά στις πολιτικές ομάδες για να υποβάλουν ερωτήσεις ή οι συντονιστές ή οι αντικαταστάτες τους. Ζων Πολ, πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Υπουργέ, εγώ θα αναφερθώ μάλλον στη μορφή και όχι στην ουσία. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ που δεχθήκατε να είσαστε ο πρώτος που συμμετάσχετε σε αυτόν τον οικονομικό διάλογο. Το ζήτησαν αυτό οι βουλευτέ. Λυπούμε που δεν είναι τόσο πολλοί αριθμοί παρόντε. Εδώ βέβαια η ποιότητα είναι την ποσότητα. Και σήμερα κατά κάποιον τρόπο μα βοηθάτε να ξεκινήσουμε κάτι το καινούριο. Δηλαδή να έρχεται κανένα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσει την κατάσταση μια οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίε και για τι οποίε η κυβέρνηση τη χώρα αναλαμβάνει κάποια μέτρα. Εγώ δεν θα ε, κρίνω κάποια από τα μέτρα σας ή να τοποθετηθώ πάνω σε κάποιους προσανατολισμούς της οικονομικής σας πολιτικής. Παρουσιάστε ένα πρόγραμμα που φαίνεται να είναι συνεπές. Μας δώσετε στοιχεία που καταδεικνύουν τη βούληση της κυβέρνησης να εφαρμόσει πράγματι τις εν λόγω προτάσεις και είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί Σκοτά σε μια έκθεση η ε, το Κοινοβούλιο έλεγε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν συνήθως τα μέτρα που εξαγγείλουν. Και τώρα η Ουγγρική ε, κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα. Ένα πράγμα θα σας πω. Σαφήλως. φοβούμαι σήμερα κάποια στοιχεία που προέρχονται από την Ουγγαρία και δεν ξέρουμε αν είναι καλά ή όχι. Και αυτό κάπως ε, ε, ε αμαυρώνει την εικόνα της ε, πολιτικής βούλησης της χώρας σας για τα οικονομικά θέματα. Και θα έλεγα ότι θα ήταν καλό το, η κυβέρνηση Ουγγαρίας, αιτήσει της Εκτελεστικής Επιτροπής, να μας δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται όσον αφορά προβλήματα που δεν είναι προβλήματα ε, οικονομικά απαραίτητο, απολυτικά και τα οποία όμως επισκιάζουν κάποια από τα μέτρα της κυβέρνησής σας, <clears throat> της οποίας την αποσυστικότητα στον οικονομικό τομέα αχαιρετίζω. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. We'll collect a few points and then and then reply uh, on behalf. Για να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις. Ξέρω σοσιαλιστών. Νομίζω ότι εσείς θα πάρετε λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξέρουμε των σοσιαλδημοκρατών της Επιτροπής εδώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο Γκοζές γιατί έχω να πω κάτι που καταδεικνύει κύριε Φουμπουργέ, το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή εδώ. Ο κύριος Γκοζές ε, το τόνισε ότι οι εντάσεις που υπάρχουν ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και της κυβέρνησης, όχι της χώρας, της Ουγγαρίας, δεν βασίζεται κυρίως σε οικονομικά θέματα, αλλά στην τήρηση προς τον ανατολισμό των ευρωπαϊκών αξιών. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί αλλού. Θέλω να το έχω πει όμως, πρωτού περάσουμε στην υπόλοιπη συζήτηση. Για να ξέρουμε και η ΜΕΝ και η ΔΕ πού υπάρχει το πρόβλημα. Του του με ενδιαφέρουν και τα θέματα τα δικά σας, τα οικονομικά θέματα. Και θα ήθελα να υποβάλω την εξή ε, ερώτηση. Σε πολλές χώρες που τις αποκαλούμε χώρες catching up που καλύπτουν το κενό, παίζει σημαντικό ρόλο το χρέος σε ε, εξωτερικό νόμισμα. Και υπάρχει το πολιτικό πρόβλημα που πώς μπορεί κανένας να το αντιμετωπίσει αυτό ως κυβέρνηση, δηλαδή πώς μπορεί με τροποποιημένους όρους ε, συναλλαγματικούς και ισοτιμιών, πώς μπορεί μια χώρα, λέω, να επιβιώσει. Με ενδιαφέρει το πρόβλημα αυτό από ουγγρικής σκοπιάς. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, τι μπορείτε να μας πείτε και όσον αφορά τις, ε, το θέμα του πόση διακριτικότητα χρειαζόσαστε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο CD4. Δηλαδή να υπάρχει μια νέα νομοθεσία για τις απαιτήσει σχετικά με τα κεφάλαια και εξετάζουμε τι θα διακανονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι σε εθνικό και ποιες θα είναι οι δυνατότητες που θα παραμένουν να οριστούν πρότυπα για τους εθνικούς επόπτες. Ευχαριστώ πολύ. So uh, uh, Σας ευχαριστώ. Πραγματικά με μεγάλη ευχαρίστηση ήρθα εδώ και εκτιμώ τα καλά σας λόγια σχετικά. Θα ήθελα να δώσω μια διευκρίνηση. Στις αγωγικέ μου παρατηρήσεις ήθελα να καταδείξω το σκεπτικό και τους λόγους γιατί κάνουμε αυτά που κάνουμε και τι κάνουμε κιόλας. Γιατί Βέβαια δεν καταλαβαίνουν όλοι στην Ουγγρική κυβέρνηση τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Αν κοιτάζει κανένας από έξω προς την Ουγγαρία δεν έχει την πλήρη εικόνα μπροστά του. Όπως είπα και προηγουμένως είχαμε επί 1,5 χρόνο μία πάρα πολύ ε, τρικυμιώδη αν θέλετε περίοδο. Εγώ θα ήθελα να σας πω τώρα βέβαια την κατεύθυνση που παίρνει η Ουγγρική ε, οικονομία. Ε, ξέρουμε από τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ότι είπε ότι ενδεχομένω θα διακόψει την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής Αρχές Φεβρουαρίου όμως, στείλαμε μια επιστολή στην Κομισιόν όπου διευκρινίσαμε τα μέτρα που θα εφαρμόζαμε κατά διάρκεια του Φεβρουαρίου για να προσαρμόσουμε τον ε, προπολογισμό μας και φέτος και του χρόνου. Και για του χρόνου οι επιπτώσεις της ε, προσαρμογής αυτής είναι 0,4%. Και αυτό έχει επιπτώσει βέβαια στο δημοσιονομικό χρέος. Το έλλειμμα μας που προβλέπει η Κομισιόν για το επόμενο έτος είναι 3,25%. Λοιπόν, 3,25 μείον 0,4 ε, πέφτουμε κάτω από το 3%. Η Ουγγρική κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να κρατήσει το έλλειμμα της κάτω από το 3%. Αυτό είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ουγγαρίας. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα μπορέσουμε να μειώσουμε σιγά σιγά το χρέος. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Να έχουμε δηλαδή το έλλειμμα κάτω από το 3%. Έχουμε ε, καθιδρύσει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να εξασφαλίσουμε ότι ο προορισμό μα θα είναι κάτω του 3% όσον αφορά το έλλειμμα το επόμενο έτο. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί και για άλλη μέτρα. Και ξαναλέω, είναι πολύ τριγυμιώδε οι εποχέ στι οποίε ζούμε. Και χρειάζεται προσαρμογή του προπολογισμού ε, στη τάξη του 4% γιατί είδαμε ποια είναι τα ποσοστά ανάπτυξη που έχουν βέβαια σημαντικέ επιπτώσεις στην Ουγγρική οικονομία. Που οπωσδήποτε έχουμε αποφασίσει να διατηρήσουμε το έλλειμμα του προπολισμού τα επόμενα χρόνια κάτω από το 3%. Κάναμε κάποιες προτάσεις ήδη το Φεβρουάριο και η Κομισιόν φαντάζομαι θα αποδεχθεί ότι αυτό έχει πραγματικά τις επιπτώσεις που αναφέρουμε. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε και είναι θέμα της εμπειρίας μας νομίζω. Ποια είναι η εμπειρία που έχουμε στην αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους ε, ή του χρέους του πληθυσμού σε ε, αλλοδαπό νόμισμα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο σίγουρα και δεν υπάρχει καμία εύκολη λύση. Δεν θα βρει κανένας κάποια εύκολη λύση. Εμείς είμαστε στην κυβέρνηση. Πρέπει να δράσουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Εξέτασα πολλές μελέτες χωρίς να βρω κάποια λύση. θα πρέπει να είναι δηλαδή εστιασμένο, η, η, κλίμακα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ουγγρική κυβέρνηση εργάστηκε επί 1,5 χρόνο περίπου και βρήκαμε νομίζω μια λύση δεχτεί για όλους. Εστιασμένη και αυτή, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα που χρησιμοποιούνται κάποια σχέδια προστασίας για εκείνους που μπορούν να τα πληρώσουν. Για εκείνους που δεν δρούν όπως θα έπρεπε, υπάρχει η δυνατότητα ε, μετατροπής του χρέους με ε, διαγραφή του 25% του χρέους αυτού. Οπότε υπάρχουν απώλειες των τραπεζών και από τις δύο πλευρές και οι τράπεζες σε αυτή την προκειμένη περίπτωση μπορούν να δια... εκπέσουν ένα 30% του ναπολιών τους. Έχουμε μια εταιρεία για τη διαχείριση των διεθνών ε, των ε, εσωτερικών οικονομικών που θα αγοράσει 25.000 σπίτια από εκείνους που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το ενυπόθηκο ε, χρέος τους. Δεν υπάρχει κάποια εύκολη λύση. Το πιο σημαντικό είναι μετά τις συμφωνίες 15 Δεκεμβρίου είναι ότι συμφωνήσαμε με τις τράπεζες. λέγοντας ότι το τέλος της τράπεζας θα μειωθεί κατά το ίμιση το 2013 και το 2014 θα έχουν εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ή Μάλιστα μπορεί να είναι και χαμηλότερο από το όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το τέλο τη τράπεζας. Πρόεδρο. κοιτάξτε, θα πάρουμε άλλε δύο ερωτήσει πάλι. Ο Σμιτ πρώτα από την Άλντε και μια που δεν έχουμε προσώπους από άλλε πολιτικέ ομάδε. η επόμενη ερώτηση θα είναι από την ε, Κάνιν Φαντικούλ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εμείς οι φιλελεύθεροι εκτιμούμε πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Εγώ έχω μια πολιτική μνήμη από το 1956 και ξέρω ότι οι Ούγγροι είναι τολμηροί άνθρωποι και γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα που έχετε έρθει. Η πρώτη μου ερώτηση είναι κάπως γενική, αλλά ελπίζω να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η Ουγγαρία τη χάνει σωστής και δικαιολογημένης μεταχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά και το θέμα των παγωμένων ποσών του ταμείου για το επόμενο έτος. Το άλλο επίσης είναι το Europlus. Εγώ είμαι από, την, από τη Σουηδία και είμαστε σε κάποιες δύσκολη θέση όσον αφορά αυτό το Europlus. Εμείς είμαστε εκτός. Νομίζω ότι είναι λάθος ε, της χώρας μου. Εσείς τι πιστεύετε για την Ουγγαρία, θα μείνετε εκτός του συμφωνίας Europlus τη σήμερα ημέρα. Και το τελευταίο η αφορά γενικά το ευρώ. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για να ενταχθείτε στο ευρώ. Ευχαριστώ. Corinne. Uh, thank you very much for being, uh, uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μας και δεδομένου ότι εσείς ε, ξεκινήσατε αυτό το πακέτο των έξι τομέων ε, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη συζήτηση για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών μέτρων στην Ένωση έτσι ώστε να μην μας κατηγορούν ότι εφαρμόζουμε αντιδημοκρατικές διαδικασίες και ότι είμαστε αδιαφανείς. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που έχετε μια ανοιχτή προσέγγιση σε αυτό το διάλογο. Όσον αφορά τώρα την, ε, την πολιτική, τις πολιτικές σας στην Ουγγαρία βεβαίως έχει άμεση σχέση με το πακέτο αυτό, τον 6. Μιλήσατε για δημοσιονομική πεισαρχία, διαρθρωτικές αλλαγές. Όλα αυτά είναι σέματα κλειδιά για την οικονομία. Ε, και είπατε, δείξατε δηλαδή ότι τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι τόσο άσχημα για το άμεσο μέλλον. Έχω όμως δύο-τρεις ερωτήσεις συγκεκριμένες που θέλω να σας θέσω. Καταρχάς, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν καλύπτει μόνο ποσοτικά στοιχεία, αλλά και ποιοτικά, την ποιοτική πλευρά των δημοσίων ε, οικονομικών. Είπατε ότι χρησιμοποιήσατε τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα εντάξατε στον ε, προϋπολογισμό για να μειώσετε το έλλειμμά σας. Αυτό, αυτή η μέθοδο δεν θεωρείται ε, ε, ε, σωστή, δεν ενδείκνυται για μια σταθερή πολιτική, για μια σταθερή ανάπτυξη και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα αν συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια. Επίσης αναφέρατε τις κυρώσεις, τις οποίες ανέφερε ήδη και ο Πίτροπος και ρωτώ τι μέτρα θα λάβετε στους ερχόμενους μήνες για να ε, ευσυγραμμίσετε τις πολιτικές σας με αυτούς κοινού ευρωπαϊκούς στόχους, σύμφωνα με αυτό το πακέτο των έξι τομέων διότι θέλουμε όλοι μας ε, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να επαναφέρουν μάλλον την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αναφέρατε την Κριστίν Λαγκάρτ και είπατε ότι ακολουθεί μία υπεύθυνη και συνετή Προσέγγισε, αλλά από ό,τι ξέρω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνείται να συμμετάσχει σε ένα, ένα πρόγραμμα στήριξης της Ουγγαρίας. Ε, πώς αντιδράσατε σε αυτό, έχετε πρόθεση να συνεχίσετε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Δέλτα Νιτάφ ή όχι, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας αυτό. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα ε, ξεκινάμε τον πραγματικά, τον ουσιώδη οικονομικό διάλογο και δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ωραία. Για την πρώτη ερώτηση, πώς, εάν θεωρώ ότι μας έχουν ε, χειριστεί δίκαια και θεμητά, αυτό μου έχουν ρωτήσει πολλές φορές τη δημοσιογράφοι, αν έχουμε τύχει δηλαδή δίκαιο χειρισμό. Όταν αντιμετωπίζουμε ελπίζω αυτή την ερώτηση ε, διαφέρει από το τι θα απαντήσει και με το τι θα πρέπει πραγματικά να, να κάνουμε στην οικονομία. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, όχι το πώς, ε, τι μεταχείριση έχουμε τύχει, αλλά τι πραγματικά κάνουμε, τι εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα, στην πραγματική οικονομική ζωή. Σας είπα ότι αυτό το ποσοστό του κάτω από 3% του προϋπολογισμού ε, δικαιολογείται, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη την οποία δέχεται και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Ε, εμείς λέμε ότι θα είναι 2,5% το έλλειμμα, η Κομισιόν λέει ότι θα είναι 2,8%. Εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε ότι θα είναι κάτω από 3%. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο και από την άλλη πλευρά επίσης ε, εξελίσσεται ένα ολόκληρο φάσμα μεταρρυθμίσεων. Και πιστεύω ότι αυτά τα, τα ρυθμιστικά μέτρα θα έχουν μια μεγάλη επίπτωση, επικοδομητική επίπτωση στην οικονομία και την αντιμετώπιση της κρίσης. Άλλο λοιπόν τι αισθάνεται κανείς και άλλο τι πράττει. Πρέπει να δράσουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε. Το Europlus, το, το σύμφωνο Europlus, εμείς είχαμε ε, συμμετάσχει όπως ε, δεν είχαμε συμμετάσχει ακριβώς όπως η Σουηδία διότι είχαμε πρόβλημα όπως την εναρμόνιση της φορολογίας. Ε, είχαμε ορισμένα καυτά θέματα στα οποία δεν συμφωνούσαμε και δεν είχαμε συμμετάσχει. Όμως, κάναμε πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, προ, κατάργηση της πρόορης συνταξιοδότησης κλπ. κλπ. στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων. Επιτελέσαμε λοιπόν και εφαρμόσαμε διάφορα μέτρα που είναι μέσα στο γύρο χωρί χωρίς να είμαστε εμείς εντός. Επίσης η Ουγγαρία και άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες θέλουν να είναι ανταγωνιστικές ε, ε, και να έχουμε την ε, εθνική κυριαρχία επί το, του δημοσιονομικού και φορολογικού πλαισίου. Ε, θέλουμε να μπορούμε εμείς ε, να αποφασίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα αυτή τη δέσμη των έξι ε, πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ουγγρικής Προεδρίας. Το πακέτο αυτό, ε, το οποίο προωθήσαμε, παρουσιάσαμε και προωθήσαμε και βεβαίως σεβόμεσα τους κανόνες αυτούς ε, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της πειθαρχίας του προϋπολογισμού. Για να μπορέσουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε χρόνο. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να μπορούμε να, να, να, μπορούμε να αγοράσουμε <laughs> αυτό το χρόνο. Ξέρω ο, και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ότι η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα αγοράζει χρόνο στηρίζοντας ορισμένα κράτη ώστε να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Εμείς όμως, συγγνώμη, ε, ε, διακόπτει η πρόεδρος, εδώ ακούγεται ο κάθε ψήσιρος η κάθε ε, συζήτηση και θα ήθελα παρακαλώ να σεβαστεί τον ομιλητή όταν μιλά και να κάνετε ησυχία. Λοιπόν, το να κερδίσουμε χρόνο και χρόνο ε, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν είμαστε μέλος της Ευρωζώνης, οπότε πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να κερδίσουμε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο. Αυτό ακριβώς ε, κάνουμε και πιστεύω ότι το εκτελούμε με πάρα πολύ σωστό τρόπο το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα. Ε, συζητάμε με το Δέλτα Νιτάφ και την Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή. Θα συζητήσουμε. Οι διαβουλεύσεις αυτές δεν άρχισαν ακόμα. Some, uh, Είμαστε εν αναμονή πρέπει, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνουμε μια προληπτική συμφωνία, να συζητήσουμε και να δούμε τέλο πάντων τι, πρέπει να γίνει πριν αρχίσουν επισήμως οι, οι τυπικές διαβουλεύσεις. Στις 17 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή ε, η Κομισιόν έστειλε επιστολή στην Ουγγαρία ρωτώντας τι θα γίνει και στις 17 Φεβρουαρίου στείλαμε εμείς απάντηση. Τώρα περιμένουμε νέα ανταπάντηση της Κομισιόν και μετά μπορούμε να αρχίσουμε τις επίσημες διαβουλεύσεις. Διότι θα πρέπει και η Κομισιόν και το ΔΕΛΤΑ και η Ουγγαρία να προχωρήσουν ταχαίως σε αυτές τις διαπραγματεύσεις η πρόεδρος. Πρέπει λίγο να επιταχύνουμε. Μετά από σε αν θα μιλήσει ο Θείοντορ και η Προβάνς και δυο το ερωτησούλες ακόμα. Μία ερώτηση διευκρινιστική. Είπατε σωστά ότι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν χρόνο και λόγω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτός ο χρόνος αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αλλά θα πρέπει και το Νιτάφ να είναι έτοιμο όταν κλεισεί ε, να βοηθήσει. Είπατε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στήριξης της Ουγγαρίας από το Νιτάφ. Ε, έτσι σωστά κατάλαβα. Αυτό που ήθελα να πω, λέει ο υπουργό είναι ότι επιτύχαμε αυτά τα οποία προτείναμε να κάνουμε, τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το, το τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν ένας χρόνος μεγάλων ανακατατάξεων και Τώρα το, το μήνυμα ε, είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λέει το Δέλτα Νιτάφ ότι πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Εμένα όμως η απόψή μου είναι διαφορετική, διότι βλέπετε το μεγάλο ποσοστό βεβαιότητας που υπάρχει στη, στην Ένωση και την Ευρωπαϊκή Αγορά, ε, η οποία βεβαιότητα έριξε την αξία των Ουγγρικών ομολόγων. Η Ουγγαρία μπορεί να βγει στην αγορά με τα ομόλογα, τα έχει κάνει στο παρελθόν και μπορεί να το κάνει και στο μέλλον. Όμως, σε ποιο επίπεδο, για, πόσα χρόνια, όταν οι αποδόσεις είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο των μέσων αυτών, των ομολόγων αυτών, είναι σημαντικότατο η Ουγγαρία να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Εάν υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, μπορεί κανείς να ε, προσφέρει χαμηλότερες απαιτήσεις, αλλά σταθερότερη συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν θέλω να αναφέρω χώρες, ορισμένες ε, νότιες χώρες, της ευρωπαϊκές, γιατί η απόδοση των ομολόγων ξεκίνησε από 7 και σήμερα είναι 3% λόγω της μεγάλης παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να υποφεληθούμε αυτή την παρέμβαση, άρα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα άλλο δίκτυο ασφαλείας. Αυτό είναι ακριβώς το δίκτυο ασφαλείας μας, το δίκτυο ασφαλείας μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι διαβουλεύσεις που θα κάνουμε. Okay, so, um... Theodore. Ευχαριστώ, Ντόρ. Ευχαριστώ. Σωστά, σωστά. Η Ουγγαρία είναι ένα ε, αναπτυγμένο ε, κράτος, αλλά όχι όσο η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες χώρες της ε, Ένωσης. Και η Ρουμανία είναι λιγότερο αναπτυγμένη από την Ουγγαρία. Καμιά φορά Αναρωτιέμαι εάν οι διεθνείς οργανισμοί, το ΔΕΛΤΑ, η ΤΑΦ και άλλοι μπορούν να διαπιστώσουν, έχουν ξεκάθαρη εικόνα των διαφορών μεταξύ των κρατών. Μελέτησα με μεγάλη προσοχή τα μέτρα της Ουγγρικής κυβέρνησης και της Ρουμανίας αντίστοιχα και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης άλλων χωρών και προσωπικά πιστεύω ότι η επιπλέον φορολόγηση διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ήταν ένα πολύ καλύτερο μέτρο από τη μείωση των μισθών. Οι γνώμες διαφέρουν βεβαίως. Ορισμένοι αναλυτές και μεταξύ των αναλυτών υπάρχουν διαφορές, διαφορά απόψεων. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας μας είπε τώρα ότι η, οι διεθνείς οργανισμοί, οι, οι πρόεδροι των τραπεζών ε, πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Ε, και ότι αυτά τα μέτρα ας πούμε θα τα λάβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως αν λαμβάνουν ένα μέτρο το οποίο δεν είναι κατάλληλο γιατί δεν μπορούμε να το επικρίνουμε. Α, μας λένε διακυβεύεται η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, της Ουγγαρίας ας πούμε ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε δεν φταίει η Ουγγαρία στα λιγότερα ανεπτυγμένα κράτη όπου η δημοκρατία βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη ε, σε αυτές τις χώρες υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τα εισοδήματα. Τα εισοδήματα των στελεχών, των ε, ε, εποπτικών οργανισμών και των οργανισμών ελέγχου η Κομισιόν είπε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε διότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία αυτών των ελεγκτικών οργανισμών χωρίς όμως να καταλαβαίνουν ότι αυτές οι νεόποπες οικονομίες οι οποίες πρόσφατα εκδημοκρατικοποιήθηκαν ισχύουν ειδικέ καταστάσεις, εξαιρετικές καταστάσεις ιδίω στη Ρουμανία. Παραδείγματος χάρη εκεί η εποπτική ε, αρχή για την ασφαλιστική αγορά. Εκεί το εισόδημα, το, η μισθή του Διοικητικού Συμβουλίου, ας πούμε, είναι μεταξύ 5 και 10 ε, χιλιάδες ευρώ, ενώ ο μισθός, το εισόδημα του Προέδρου της Δημόσιας Υπηρεσίας για τον Έλεγχο των Ασφαλιστικών Εταιριών είναι 27.000 ευρώ. Και ο μέσος μισθός στη Ρουμανία είναι 500 ευρώ. Προσέξτε. Η θέση της Κομισιόν και του Δέλτα Νιτάφ μας είπε μην, μπλέκε, εμπλακείτε σε, αυτό, αυτή τη συζήτηση, είναι θέμα ανεξαρτησίας των φορέων αυτών. Ε, μην παρεμβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να υπεραμεινθεί τέτοιων ε, αποφάσεων, μια τέτοια κατάσταση η Ουγγαρία έναντι της, της τράπεζα Τράπεζας και του ΔΕΛΤΑ Η Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Υπουργέ. Καταρχήν η χώρα σας είναι η πρώτη που υποφελήθηκε από τη διευκόλυνση του ισοζυγίου πληρωμών. Δεν ήσασταν τότε υπουργό, αλλά όταν φτώσατε στην εξουσία η κατάσταση ε, βρισκόταν σε εξέλιξη. Τι κάνατε λοιπόν ε, με αυτή τη διευκόλυνση που χορηγήθηκε στην χώρα σας. Δεν έχω την εντύπωση ότι η διαχείριση αυτής της διευκόλυνσης επέτρεψε να αποκαταστησετε την κατάσταση. Είπατε ότι πάμε, προχωράμε γρήγορα, υιοθετήσαμε πάνω από 300 κείμενα, αλλά μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποια ασυμβίβαστα με το ευρωπαϊκό πνεύμα και ειδικά το ζήτημα της εξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν αφισβητώ πως ε, σε επίπεδο αμοιβών μπορεί να υπάρχουν κάποιες υπερβολές σε σχέση με το μέσο μισθό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δίνεται στην Κεντρική Τράπεζα και αναφέρατε το ζήτημα της σημασίας της ε, ζώνης ευρώ και την συνέργεια που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη ζώνης ευρώ και μη μελών αυτής, κάτι που δεν αφισβητώ αλλά στην περίπτωση αυτή το καθεστώς της τράπεζας σας και η συνθήκε μέσα στι οποίε προετοιμάζεται να γίνετε ένα πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν στιγματίζετε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει και μεταχειρίζεται την ε, Ουγγαρία. Κοιτάξτε, δεν νομίζω πω η ε, ε, Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αποτελέσουν τον αποδιομπέο τράγο σε πλαίσιο τη ιστορικής σας και βλέπω ότι δεν, ε, ε, ότι δεν φροντίζεται να ε, προσφέρετε να δώσετε τις κατάλληλες απαντήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κομισιόν. Όταν λέτε ότι υιοθετήσατε χ κείμενα, πείτε μου με ποιο τρόπο τα κείμενα αυτά διευκόλυναν αυτό, αυτούς που, αυτό που στην χώρα σας ε, ευνοούν και δει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον ε, οικονομικό ιστό. Μου λένε ότι η κατάσταση σε αυτές τις επιχειρήσεις έχει επιδεινωθεί λόγω της γραφειοκρατίας ε, που εφαρμόζεται και τα μέτρα γραφειοκρατικά που λάβατε. Τι κάνετε τώρα σε θέματα φορολογίας, διότι μία από τις δυσκολίες ε, της χώρας σας νομίζω είναι ακριβώς η φύση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που εισάγατε. Εγώ δεν ε, υποστηρίζω το Pact Plus, ε, δεν είναι... Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να το δεχτείτε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν σωστό να το πράξετε, να δεχτείτε αυτό το σύμφωνο. Υπάρχουν μια σειρά από ανισότητες, ειδικά στην αγορά εργασίας και θα μπορούσατε να είστε ένα πολύ καλό, θα μπορούσατε να είστε ένα, πολύ καλό παράδειγμα, κάτι όμως το οποίο δεν το πράξατε τώρα για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Πώς πιστεύετε ότι αδειώσει τα πράγματα για να υπάρξει χρηματοδότηση του χρέους σας παρά να επιδεινώνετε τις ανισότητες όπως συμβαίνει μέσω της, του καταποκοπήν φόρου, καταποκοπή τέλους που εισάγατε. Και τέλος ε, αναφέρεστε σε αποτελέσματα τα οποία και διεκδικείτε. Ε, αλλά όλοι γνωρίζουν πώς πετύχατε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι ε, Πρόκειται για μια επιχείρηση one shot, ε, δηλαδή μεταφέρατε τα κονδύλια των ε, Ταμείων Συνταξιοδότης. Πώς θα ακολουθήσετε λοιπόν αυτήν την ε, στρατηγική, διότι δεν υπάρχουν πολλά ιδιωτικά ταμεία, τα οποία συνταξιοδοτικά, τα οποία θα μπορούσατε να μεταφέρετε στον ε, κρατικό προπολογισμό. Um, we haven't got a great deal of time. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε δύο ερωτήσεις γιατί ο Υπουργός θα απαντήσει ομού με όλες. Σίλβη, Σίλβη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που... Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Χαιρόμαστε που δεχθήκατε. Εμεί είμαστε εξάλλου και εισηγητέ ε, του Six Pack. Ευχαριστώ και του όγκρου ε, ε, αξιωματούχου που μας βοήθησαν σε αυτό το πακέτο. Μια γενική, γενικότερη ερώτηση με ειλικρίνεια. Δεν έχει την εντύπωση ότι η μεγαλύτερη αξία που συμμεριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σεβασμός του δικαίου. Και ο σεβασμός ενός κράτους δικαίου επιτρέπει στον πολίτες να ζουν ε, ορθά, αλλά και στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εργαστούν. Στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας, τα ερωτήματα που αφορούν στις ασφαλιστικές εταιρείε ε, σε όλοι όσοι υπέστησαν βίες ε, νομοθετικές αλλαγές δεν έχετε εντύπωση ότι όλα αυτά θα περιπλέξουν την κατάσταση σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πλήξουν και την εικόνα της Ουγγαρίας. Δεν μιλάω ε, λόγους ιδεολογικούς. Ε, αν κάποιος θέλει να επενδύσει τη χώρα σας έχει την εντύπωση ότι οι συμβάσεις θα τηρηθούν, ότι έχει να κάνει με θεσμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα που είναι ανεξάρτητη. Με λίγα λόγια λοιπόν, παραμένετε στον ευρωπαϊκό δρόμο, στην ευρωπαϊκή οδό, θέλετε να φτάσετε κάποια στιγμή στο ευρώ, όπως ρώτησε και ο κύριος Σμίτου. Νομίζω ότι υπάρχουν δεσμεύσει και θα πρέπει να τις σεβαστείτε, να τις στηρίσετε και να τις κάνετε δικέ σας. Τα λέω όλα αυτά προερχόμενα από μια χώρα που δεν ήταν ε, υποδειγματική στην τήρηση των ε, οδηγιών. Δεν θέλω να σας πετάξω κανένα μπαλάκι. Ε, θεωρείτε λοιπόν ότι η στάση σας είναι κατάλληλη ή θα πρέπει να σεβόμαστε όλοι το κράτος δικαίου. Τελική ερώτηση, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υφυπουργό και την παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την, ε, τις άνετες απαντήσεις ε, που έδωσε μέχρι τώρα, αλλά όχι και πάντα στις ε, ερωτήσεις. Είμαι μέλος του κυβερνώντος κόμματος στην Ουγγαρία. Πρέπει λοιπόν να δεχθείτε την θέση μου ε, ε, ως αντικειμενική. Είμαι οικονομολόγος, ε, πιστεύω στους αριθμούς και πιστεύω επίσης πως τόσο η Κομισιόν όσο και εσείς μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτά τα, στους αριθμούς χωρίς προκατάληψεις. Όταν η Ουγγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η διαδικασία ε, υπερβολικού ελλείμματος ξεκίνησε και τότε το έλλειμμα ήταν μεταξύ 6 και 9% για μερικά χρόνια. Μια χώρα η οποία δεν ε, είχε καμία οικονομική ανάπτυξη, σε ένα χρόνο ε, το ΑΕΠ της Ουγγαρίας μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα που ακόμα πριν από την κρίση έπρεπε να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να της χορηγηθεί ε, δημοσιονομική υποστήριξη και αν δεν της είχε δοθεί τότε η Ουγγαρία θα είχε πτωχεύσει. Ουγγαρία όμως ε, μετά ακολούθησε μια περίοδο ύφεση ε, όταν ε, άλλαξε η κυβέρνηση στην Ουγγαρία το 2010. Τώρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έδειξε μάλλον η οποία συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μείωσε το έλλειμμα. Παράλληλα ξεκίνησε προσπάθειες ανάπτυξης και ανάκαμψης. Η Κομισιόν εξετίμησε αυτή την ε, επιθυμία της ε, Ουγγαρίας ε, μειώθηκε το έλλειμμα της Ουγγαρίας πέρυσι, η οικονομική ανάπτυξη ήταν στα 1% και η Κομισιόν λέει ότι δεν είναι τα μέτρα που δεν της αρέσουν, αλλά είναι το πνεύμα που δεν αρέσει. Δεν το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι τα στοιχεία, οι αριθμοί. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει η οικονομία είναι καλή και οι στόχοι της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης είναι και αυτοί ικανοποιητικοί. Ναι και θα θέλω να θέσω τώρα την ερώτηση Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα δρατώ με τις ευκαιρίες... Ε, να πω και κάτι γενικότερα στην Επιτροπή μας. Έχω μια ερώτηση όχι μόνο προς τον Υπουργό, αλλά και προς τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι καλά, αλλά η Κομισιόν ε, συνεχίζει να δηλώνει ότι η στάση της κυβέρνησης δεν είναι η κατάλληλη, διότι τα μέτρα... Κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε. Αν ε, πιστεύετε στους αριθμούς και στα στοιχεία και αν ε, είστε ικανοποιημένοι με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε, τι θεωρείτε απαράδεκτο. Έχω την εντύπωση πως ε, η Ουγγαρία Κοιτάξτε, πρόκειται για έναν οικονομικό διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και τον Ούγγρο Υπουργό. Και επί και σας ακούσαμε τέσσερα λεπτά και τώρα δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε τον ε, Υπουργό. Έχετε κάποια ερώτηση προς τον Υπουργό, λυπάμαι, αλλά κοιτάξτε πως ο χρόνος τρέχει και εσείς ερώτηση δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ήδη έθεσα ερώτηση με, στην τελευταία πρόταση και λυπάμαι που σας τεραχωρήσα. Πρόεδρο. Έχω λίγο χρόνο. Γκοζέ, πρόεδρε, εάν θέλετε τάξη πρέπει να θέσετε τάξη στο σώμα. Λοιπόν, οι επισκέπτες που βγαίνουν για να κάνουν τη βόλτα τους δεν πρέπει να κάνουν θόρυβο. Θα θέλουμε να ακούσουμε τον Υπουργό και να υπάρχει πλήρης σιωπή. Δεν είναι σαλόνι για να κάνουμε κουτσομπολιά. Η Επιτροπή μας ε, Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Θα φροντίσω να είμαι σύμφωνο, σύντομος σύμφωνα με την νομοθεσία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας είναι ανεξάρτητη, ήταν και θα είναι. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Και κοιτάξτε, όχι επειδή κάποιος το ζητάει, αλλά διότι η εμπειρία μας μας λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη για να ελέγχει την εξέλιξη των τιμών και τη σταθερότητα. Πρόεδρος, παρακαλώ, ψήθυροι ακούγονται μέχρι εδώ πάνω. Εγώ μεταβίας ακούω τον κύριο Υπουργό όταν μιλάει. Παρακαλώ, σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας ή με οποιονδήποτε άλλον δεν πρόκειται να ξεκινήσει η συνεδρίαση εάν δεν σιωπήσετε. Στα μέσα του 90 λοιπόν στην Ουγγαρία είχαμε ε, πληθωρισμό 25-27% για δύο χρόνια. Ξέρουμε πόσο επίπονο είναι κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον των 10 εκατομμυρίων των Ούγγρων η τράπεζά τους η κεντρική να είναι ανεξάρτητη και να συνεχίσει να παραμένει ανεξάρτητη έχει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για θέματα πληθωρισμού και σταθερότητα των τιμών. Τώρα για την ε, θέμα της παραβίασης ε, η Κομισιόν έθεσε έξι ερωτήσεις, ε, εκκρεμούν δύο απαντήσεις με οποίες, για τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτούμε ακόμα. Το ένα αφορά ότι ο κυβερνήτης, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να ε, από κάποιους κανόνες και Υπάρχει και το θέμα της, ε, του συντάγματος αλλά και της τήρησης ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εδώ γίνεται αναφορά και στην ανεξαρτησία. Again, Πάλι συνεχίζετε να ομιλείτε και να κάνετε κουσκούς. Επίσης ε, έχει τεθεί το ζήτημα του διοικητή, όπως σας είπα, της Κεντρικής Τράπεζας και των ε, υπολείπων ε, αξιωματούχων, και για αυτούς θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες. Η Κομισιόν είπα, έθεσε έξι ερωτήματα, σε τέσσερα ζητήματα εμείς δεχτήκαμε τις θέσεις τους, όπως το ζήτημα της συγχώνευσης κάποιων ε, οργανισμών και υπάρχουν δύο θέματα που εκκρεμούν αλλά μπορούμε εντάχει να τα διαπραγματευτούμε και αυτό δεν φύγει ε, την εξαρτησία της κεντρικής του τράπεζας διότι όπως προείπα είναι προς το συμφέρον 10 εκατομμυρίων Ούγγρων ε, η κεντρική μας τράπεζα να είναι και να παραμείνει ανεξάρτητη. Τώρα για τον αποδιοπηπαίο τράγο που είπατε, αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Στην οικονομική πολιτική πρέπει να κάνουμε το, το έργο μας, το καθήκον μας και αυτό έχει σημασία. Πρέπει να καταρτήσουμε ένα προπολογισμό, πρέπει να μειώσουμε το χρέος και αυτό κάνουμε. Τώρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις προωθούμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις ε, για τις μικρές επιχειρήσεις. Να αναφέρω ένα στοιχείο. Χθες ανήγγειλα ότι στην Ουγγαρία με τη στήριξη των διαχωρικών ταμείων ε, και των ε, ταμείων που διαθέτουμε τη χώρα θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη και ένα μεγάλο ποσοστό θα δοθεί στι μικρές επιχειρήσει Τώρα για το διοικητικό άχθος, ένα στοιχείο. Μειώσαμε κατά 50% αυτό το άχθος. 600, 600 ε, διαφορετικές ρυθμίσεις ίσιαν πριν αναλάβουμε εμεί και τώρα μειώσαμε στο 50%, δηλαδή υπάρχουν 300 τώρα το συμμετοχή στο στο ευρώ. Πρώτα όμως, πρώτα πριν συμβεί αυτό θα πρέπει να πληρούμε τις ε, προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε, τις οποίες έχουμε προσυπογράψει. Το πρόβλημα μας είναι το χρέος, ε, το οποίο δεν είναι κάτω από 80%. Χρειαζόμαστε όμως για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το ποσοστό αυτό μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και φυσικά το έλλειμμα του προβλησμού πρέπει να είναι 30%. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να ενταχθούμε στο ευρώ. Πρώτα θα πρέπει να πληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις το πυλώνας ε, των ε, ε, ιδιωτικών συντάξεων. Χρησιμοποιείτε τη σωστή ορολογία. Mandatory, υποχρεωτική, δεσμευτική. Πώς μπορεί να είναι κάτι ιδιωτικό όταν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει εδώ ένας αλληλογροθοσκοπισμός των δύο αυτών Τι είδους αγορά έχουμε όταν έχετε τέτοια θεσμού, τέτοιου φορεί ε, σε εξωτερικού, ε, πώ μπορείτε να ανταγωνιστείτε στην αγορά όταν ε, ο, ο πολίτη είναι υποχρεωμένο, όταν έχουμε mandatory συμμετοχή. Κάθε χρόνο στον προπολογισμό είχαμε μια τρύπα 1,4-1,5%. Γιατί η Ουγγαρία είχε αυτή την αύξηση του χρέους. Ένας λόγος ήταν ακριβώς αυτός. Πρόκειται για έναν ε, προαιρετικό, εθελούσιο προαιρετικό πυλώνα και όχι υποχρεωτικό. Τώρα, τα στοιχεία να αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Το 2002, εκλογική χρονιά, είχαμε 9% έλλειμμα. Το 2016. Το 2010 είναι η πρώτη χρονιά όπου μπορέσαμε να βελτιώσουμε τον προπολογισμό και το 2010 είχαμε ένα ε, το 2011 είχαμε ένα έλλειμμα κάτω του 30% και φέτος ε, νομίζω ότι θα το πετύχουμε πάλι και νομίζω αυτός είναι σωστός τρόπος ε, για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε μεταξύ μας. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, αυτή η αίθουσα είναι προβληματική για να έχουμε συνεδρίαση και ειδικά με πολλούς παρόντες. Ε, Ακούγονται, έχει πολύ ηχό. Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της μεσης ε, ψυχοφορίες. Σας ε, αφήνω μερικά λεπτά για να κοιτάξετε τον κατάλογο των ψηφοφοριών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 Okay, could everybody take their seats, please? Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σα. Έχουμε αρκετή δουλειά. Το κακό είναι ότι θα πρέπει να ακούσετε και τι ανακοινώσει του Προέδρου που είχαν αναβληθεί μέχρι τώρα, γιατί είχαμε καθυστέρηση με το χρονοδιάγραμμά μα. Πρώτον, θα πρέπει να σα πω ότι πήγε μία αντιπροσωπή τη ΕΚΟΝ στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κόνγκ την περασμένη εβδομάδα. εγώ, Μπροτοθόλη και η Αλμακάρθη είχαμε συναντήσει καταρχήν στην Πακούρη με υπουργού και υφυπουργού ε, οικονομικών, με τον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου και με τους επικεφαλείς ε, του χρηματιστηρίου, την Ένωση των Μετοχών και Επενδύσεων και την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Στο Χονγκ Κόνγκ με τον Υφυπουργό για Οικονομικές ε, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, πρόεδρο του Συμβουλίου, του Νομοθετικού Συμβουλίου, του Χρηματοστηρίου, τη Επιτροπή των ε, Μετοχών και Ένωση ε, των Τραπεζών και του προγράμματο ενημέρωση επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε χρηματοπιστωτικά θέματα, ταυτόχρονα όμω, ε, εξετάσαμε το θέμα τη ε, κρίση του ευρώ και πολλά άλλα, μεταξύ των οποίων και το θέμα των ε, εξοχρηματιστηριακών παραγόγων. Όπω σα είπα, το κρατικό χρέος επίσης και του θέματο του ευρώ και μαζέψαμε πολλές χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για δική μα νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής του 2012 γιατί μετά από μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια υπάρχουν ε, αλλαγές ε, στο προπολογισμό και δεν μπορούμε να έχουμε συνεδρία στην Τρίτη και Τετάρτη μόνο. Πρέπει να έχουμε ή Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη, Πέμπτη. Αναγκάσαμε λοιπόν να μεταφέρουμε κάποιες ημέρε συνεδρίασης. Και λόγω του βεβαρημένου προγράμματος εργασία της Επιτροπής μας, οι συνομιστέ αποφάσισαν ότι θα ήταν καλό να ειδοποιήσουμε την διοίκηση ότι στις 15, 23, 39 και 49 εβδομάδες θα χρειαστούμε συμπληρωματικές συνεδριάσεις. Υπάρχει επίσης και η δημοσίευση στο ιστοσελίδα της Επιτροπής των εργασιών που βρίσκονται εν εξελίξη. Μπορείτε να βρείτε αυτά στην ιστορία από την βάση δεδομένου του ΙΤΑ που χρησιμοποιείται από την γραμματεία της ε, Ολομέλειας και θα σας ε, φανεί σίγουρα χρήσιμο αυτό. Ε, θα μπορείτε να δείτε ε, ποιες είναι οι επιτουσίας αρμόδιες επιτροπές, οι, ε, οι επιτροπές που γνωμοδοτούν, οι συγητές και όδες συγητές και οι, τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι δημόσια διαθέσιμο λοιπόν στο ιστοσελίδα. Τώρα ίσως οι, οι, οι πολίτες δεν θα υποβάλουν τόσες ξεχωριστές ερωτήσεις στους συγητές και στους Επίσης σήμερα το απόγευμα η συνεδρία θα αρχίσει στις 3.30 όχι στις 3. Θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω και το πρώτο σημείο θα είναι... Όχι. Όχι, όχι, εντάξει, ωραία. Θα πρέπει να ελέγξουμε τώρα τις ε, κάρτες ψηφοφορίας. Και αν έχω πει κάτι το σφαλμένο, πως θα το διορθώσω. Okay, the, the test vote's open. Press your... Άκτη ψηφοφορία λοιπόν, δοκιμαστική. Right, we've got uh, two, two too many EPP. Δύο ΕΛΚ περισσότεροι από ό,τι χρειάζεται. Too many EPP, one too many EPP. Ένας περισσότερος, τον εντάξει. 44 κάρτες έχουν βγει, 43 ε, ε, κουμπιά όμως έχουν ε, παθηθεί. Δεν ξέρω, κάποιος έχει ξεχάσει να πατήσει το κουμπάκι. Α, τώρα έχουμε 44 με 44. Πολύ ωραία. Όλες οι μηχανές λοιπόν λειτουργούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We now start with the, um, I'll take my specs off, the draft, the draft report. Τώρα έχουμε την ε, την ε, πρόταση της κυρίας Λούνη για τραπέζι οδηγίας συμβουλίου. Συμβασμική κάπα. Α, όχι. Έχουμε πρώτα την πρόταση για απόρριψη. Πρόταση για απόρριψη του συνόλου. Άμα αυτό γίνει δεκτό, εντάξει, τελείωσε. Μπήκατε στον περασμό. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Mm. Δυστυχώς απερίφθη. Συμβαστική κάπα. Ένα τμήμα. Ναι, όλα μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 108. Υπέρ της 108, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 112, όχι, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δέκα από την τραν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι ενεκρίθη. Για να ελέγξουμε. Everybody's voted. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Πράγματι απερίφθη. Καλά που το έλεγξα δηλαδή. 20 υπέρ, 24 κατά. Εδώ 15 χρειάζεται. 7 ήτρε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 εγκρί υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 8 υπέρ, κατά, αποχές. MV16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 119 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε 119 Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Ναι. 24 υπέρ και 17 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Εννέα ήτρε υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε και αυτό. Πέρας. Α, εκκρίνεται 23 προς 9. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε να ελέγξουμε καμιά φορά είναι δύσκολο Everybody voted. Oh, right. that is actually... Ναι, πραγματικά είναι κρίθη 23 προς 21. 121 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 122 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται α να ελέγξουμε να ελέγξουμε Uh, Wait. Four, four, four more people still to vote if you're voting. Τέσσερις δεν έχουν ακόμα ψηφίσει. Ευχαριστώ. 21 προς 21. Απορρίπτεται λοιπόν, πράγματι. 125, 126 και 11 ήτρε υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε και αυτό. Everybody's voted. That's 21. 21 προς 21. Και αυτό λοιπόν απορρίπτεται. Συμβιβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Άστριτ. Μα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω κάτι για τη συμβαστική αυτή τροπολογία. Εγώ ήμουνα υπέρ της διαγραφής της αναλογικότητας που ε, απερίφθη 21 προς 21. Μέχρι σήμερα το πρωί υπήρχε όμως αυτή η συμβαστική τροπολογία L που πρότεινε 2028 για την εισαγωγή της αναλογικότητας αυτή. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλαξε αυτό και έγινε 2025. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω στους συναδέλφους να καταψηφίσουν την αυτή συμβαστική λύση και να ψηφίσουν υπέρ των τροπολογιών 127 και 128. Φίλιπ Ντεμπάκερ και Ροβάνα Πλάμπ. 128-129. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την ΕΛ. Ακούσατε την εισηγήτρια. Uh, four more people to vote, one more person to vote. Ψήφισαν όλοι πέρα ψηφοφορίες εγκρίνεται 24 προς 20 και περνάμε στην 130 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Wait, this is 130. Στην 130, την 130 ψηφίζουμε. Uh, has Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. 10-22. 131 υπέρ. Μα δεν είναι κρίθη 130. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένφι 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV19 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ Two more 23 προς 21, εγκρίνεται, 134 υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε και αυτό. Απορρίπτεται. 17 προς 21. Ήτρε 12 υπέρ. Α, είναι το ίδιο. Α, οκ, okay, οκ. 135 υπέρ. 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία μη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική νη, υπέρ, κατά, αποχές, για να το ελέγξουμε. Compromise N. N. Συμβαστική νη. Ναι. Everybody voted, votes closed. Ψήφισαν όλοι. 23 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ή 315 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 147, όχι. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 11 τραν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV20 το ίδιο 149 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε να το ελέγξουμε όμως καλύτερα Thank you. 23 in favor and 21 against. carried. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 12 τραν υπέρ, κατά, αποχές. NV21 υπέρ, κατά, αποχές. απορρίπτεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν θέλετε να ελέγξουμε, αλλά νομίζω ότι είναι κρίθη. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 χωρίς ψηφοφορία. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές να αλλάξουμε Λοιπόν, 23 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174. 173, okay. Θέλετε να ελέγξουμε την 174. Ένας ακόμα. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Ε, συμβιβασμός ε, ρο. Δεκτός. 176 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α. Λυπάμαι, Χωσέ. Συμβιβαστική. Α, δεν μπορούμε να τον επηρεάσουμε, έχει καινούρια θέσκη. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, S, S, α, S. Ναι, ναι, S. Είτε 20 υπέρ κατά αποχές Νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε την 20. 20 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή, δεκτή. 23 προς 21. 184 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 184. Ψηφίσατε, έληξε ψηφοφορία. Απορρίπτεται ξεκάθαρα. Ήτρα 21, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ένβη 25 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ήτρα 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186, 187 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 188 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 189. Απορρίπτεται 190 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 8, ε, άγκρι 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ήτρα 23 υπέρ κατά απορρίπτεται, άγκρι 9 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι μπορεί, μπορεί και να πέρασε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται, παρακαλώ. Δύο ακόμα λοιπόν, παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέραση τη ψηφοφορίας. Έγινε δεκτή, δεκτή. 27 προς 16. συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Άργησε λίγο να ψηφίσει το ΕΛΚ. 194 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, budget 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η προηγούμενη ήταν 195, συγγνώμη. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να ελέγξουμε την 199 παρακαλώ Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 29 προ 15. Ήτρα 25 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ή 200 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρα 26 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική U υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην Ήτρα 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είτε 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είτε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απορρίπτεται, ήτρε 33 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται, η 218 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική α. Α, λισό, συγγνώμη, παραλείψαμε την 22. 22 υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε τροπολογία 22 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι δύο κόμμα. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 23 προς 19. Συμβιβαστική Α. Ε, δεκτή. δεκτή. Τραν 1. Ε, υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Ενβι. 2. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 2. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές. Πιστεύω ότι απερίφθη, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Την 4 του εισηγητή. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 19 προς 24. 27 ε, ε, πέρασε, 28 απορρίπτεται, 3 απορρίπτεται, η budget 1 υπέρ κατά αποχές δε, δεκτή. Η budget 1, θέλετε να την ελέγξουμε, budget 1. Έληξε η ψηφοφορία. Α, τώρα περίφθη. Μάλιστα, μάλιστα. Περίφθη, η budget 1. Κάποιο. κάτι ήξερε ότι δεν πάει καλά. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Ποια να ελέγξουμε θέλετε. 32 μάλιστα. Την 32. Ψηφίσατε, έλεξε. Για να ελέγξουμε. 27 προς 16. Λοιπόν, προχωράμε. 34. Υπέρ, κατά, αποχές. 34 παρακαλώ, ανα, ανατάσσεως της χειρός. 34. Α, ελέγχουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πιο σίγουρα. Δεκτή, δεκτή. 21 προς 20. Ίσα ίσα. Δεκτή 34. Αγκρί 1. Υπέρ αποχές. Δεκτή. NV5. Υπέρ κατά Δεκτή. Ε, συμβιβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 6 ε, του, του, του, της ε, του Δεκτή. Για να ελέγξουμε παρακαλώ την 6 του εισηγητή, της, της εισηγήτριας. So it probably changed, but no, that is rejected. Απερίφθη, απερίφθη για μία ψήφο παρακαλώ, 21 προς 22. Προχωρούμε, 40, υπέρ κατά αποχές, δεκτή, 41 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται, 7, 7 ε, υπέρ κατά, αποχές. Νομίζω ότι λείπει μια ολόκληρη ομάδα. Να ε, ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. 7 και 43 λέει η πρόεδρος. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Α, 44 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 44. Τι έγινε με το ΕΛΚ. Ξανά παρακαλώ τη 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV6 υπέρ κατά αποχές. Ε, δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. «24 υπέρ, 20 κατά, δεκτή. Ήτρε 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 50. Ψηφίσατε, έληξε. 22 προς 22 καταπίπτει. Ένα λεπτό, διαδικαστικό. Πρόεδρε, μόλις αντελήφθη μια αποχώρηση από την ομάδα του ΕΛΚ, δεν με εκπλήσει, αλλά το διαπιστώνω. Και θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν ε, αν υπάρχει ικανό αριθμό ε, το ΕΛΚ ή αν υπάρχει κάποιο περσεκούμ που θα μπορούσε να ψηφίσει στη θέση τη απούσα. Έχουμε 44 ψήφους ε, για 44 δικαιούχους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγγνώμη για την διακοπή που οφείλεται σε κάποιες ε, αναταραχές εγώ ξέρω ακριβώς πόσοι δικαιούνται, πόσοι ψήφισαν. Οπότε ε, έχω ε, λίγο χάσει το, τον ήρμό. Εδώ είμαστε στην 50, NV7. Α. Η 50 κατέπεσε. Είμαστε στην NV7. NV7. Υπέρ, κατά απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός C ε, γάμα υπέρ κατά αποχές δεκτός ε, ε, συμβιβασμός δέλτα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ το, τη συμβιβαστική δέλτα D πέρας έληξε ψηφοφορία Καταπίπτει 22 προς 22. Τώρα πάμε στην 57. Υπέρ 57, διότι κατέπεσε η συμβιβαστική, δεν ψηφίστηκε η συμβιβαστική δέλτα, οπότε έχουμε την 57 του Μπέρντ Λάγκε. Υπερκατάποχες δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά Α, κα... πρέπει να πάμε στην 62. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική ε, ή υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Εξήντα οχτώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 Α, 70 δεν 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για να ελέγξουμε την 73 παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. 23 προς 21, άρα ε, ε, ισχύει. Πέρασε. Δεκτή. Το ε, 74 δεκτή. Το 6 ε, δεν πέρασε. Συμβιβαστική F δεκτή. Ε, συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κα, κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την συμβαστική H. Δεκτή 23 ε, προς 21. 88 υπέρ κατά αποχές. Πιστεύω ότι απερίφθη, αλλά να ελέγξουμε την 88 παρακαλώ. Παρακαλώ, ε, τρεις ακόμα, γρήγορα, γιατί έληξε η ψηφοφορία. 24 προς 20, δεκτή. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αγκρί 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ένδυ 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, Ι. Άι. Παρέλειψα τίποτα. Συμβιβαστική Ι. Άι. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αγκρι 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 95. Α, ελέγχουμε την 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευτυχώς που η Άστριτε έχει το νου της. Ένας ακόμα, παρακαλώ να ψηφίσει. Εντάξει. Έληξε η ψηφοφορία. 22-22 καταπίπτει. Πάει τώρα. Δεν πέρασε η 95. Άγκρι 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική J υπέρ... Α, πάλι χα... ε, ξέχασα την 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πριν ε, ψηφίσουμε κάνουμε την τελική ψηφοφορία θα ήθελα απλώς να ελέγξω εάν παραλείψαμε κάτι, ξεχάσαμε κάτι ε, έτσι, κάτι με, Είχα μια υποψία, αλλά όλα είναι εντάξει. Ψηφίζουμε το τροποποιησέν κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι το κείμενο όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ. Έληξε ψηφοφορία. 22 υπέρ. 6 κατά. 16 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας ακόμα, μία ψήφος ακόμα. Έληξε ψηφοφορία. 22 υπέρ, 6 κατά. 16 εποχές. Πάλι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. And congratulations to Astrid. Και συγχαρητήρια στην Astrid. One Okay, let's travel. Let's let's let's continue. Um, Συνεχίζουμε. Ησυχία στην αίθουσα παρακαλώ. Περνάμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ΚΑΖΑ για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απο, ε, δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 29 έχει αποσύρθει 30 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα ας ελέγξουμε λοιπόν 30 ε, προπολογία δεν ήμουν σίγουρη το αποτέλεσμα λοιπόν 42 ψηφι υπέρ καμία ψήφος κατά. Ε, οι μισές ε, ψήφοι υπέρ ε, έγιναν όταν είχα πει ήδη το κατά. Λοιπόν, 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 34 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 35 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 36 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 1, 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8, υπέρ κατά αποχές δεκτή 9, υπέρ κατά αποχές δεκτή 10, με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 11, υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή Το ψηφίζουμε ηλεκτρονικός επί της τροποποιηθής σας έκθεσης. Ακόμα τρεις απομένουν να ψηφίσουν. 43 ψήφοι υπέρ, Καμία ψήφος κατά, καμία από εκεί. Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα μορφωτικού περιεχομένου, την ψηφοφορία. Ακόμα έξι απομένουν. Άντε, βιαστείτε λίγο. 38 ψήφισαν, κλείνει την ψηφοφορία. 39 39 ψήφισαν, 38 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα περνάμε στην γνωμοδότηση της Έλενα Μπασέσκου. Σωσία. Ε, σας λίγο μάθαμε καμία παρα... παρατήρηση να πω στου αδέλφους ότι η ομάδα μου στην τροπολογία 20 απήχε και αυτό διότι σε συνόηση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αποφασίσαμε πως χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο να εξετάσουμε το ζήτημα διότι ε, η Κομισιόν αρχικά είπε άμεσα αυτό σημαίνει το on you delay, αλλά θέλαμε να το διευκρινίσουμε. Η Επιτροπή όμως η αρμόδια ενέκρινε την έκθεση. Εμείς ε, θέλουμε να εξετάσουμε ποιες θα είναι η επιπτώσεις αυτή την τροπολογία για την πολύ καλή έκθεση της συναδέλφου. Ευχαριστώ. Τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε ομού όλες ομαδικά, όλες τροπολογίες ε, πρόεδρα. Εντάξει, από 2 έως 14 ψήφι υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνονται. Τροπολογία 32, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 15 έως 19, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Χαρακτηριστικός μικροφώνου, ναι, γλωσσικέ φύσει ήταν αυτέ, 35 υπέρ κατά αποχές, 36 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Μπορούμε να περάσουμε στις επόμενες ομπλοκ ε, ε, λοιπόν, 15 έως 18 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός επί του συνόλου. Ψήφισαν άπαντες. Μη φεύγετε παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίστε. Έληξε η ψηφοφορία. 34 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ. <laughs>